Okay. Hello everybody. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω στη συνεδρίαση. Όπως πάντα θα μιλήσω σουηδικά. If you don't know what I'm saying, of course. <laughs> Vi eh, har här en, en stund som vi... Λοιπόν, έχουμε τώρα κάποιο χρόνο στη διάθεσή μας για να ακούσουμε τα όσα έχει να μας πει η ιδανική Προεδρία. Έχουμε τον Υπουργό για την Ισότητα των Φύλων και την Υπουργό αφασχόλησης. Θα μας παρουσιάσουν το πρόγραμμα της Προεδρίας, θα μπορείτε μετά να υποβάλλετε ερωτήσεις και θα πάτε σε απαντήσεις βέβαια. Καταρχής θα ήθελα να χαιρετήσω εγκαρδιότατα την Προεδρία εδώ μεταξύ μας, Καλωσορίσατε. ορίσατε. Θα ε, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να ακούσουμε το πρόγραμμα σας στον τομέα που μας απασχολεί. Και βέβαια ελπίζουμε ότι κατά τη διάρκεια Προεδρίας θα μπορούμε να έχουμε έναν καλό διάλογο. Περιμένουμε να ακούσουμε τι θα μας πείτε. Ο κύριος Σαρέν έχει το λόγο πρώτος. Members of the committee, Mr. Chair, I'm delighted to have uh, Κυρίες και κύριοι μέλη της Επιτροπής, κύριε Πρόεδρε, με χαρά έρχομαι να σας μιλήσω σήμερα και με χαρά θα σας παρουσιάσω τις προτεραιότητες στον χώρο των αρμοδιοτήτων μου στην ε, Προεδρία της Δανίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να αλλάξουμε απόψεις ώστε να έχουμε μια πλήρη και επικοδομητική συνεργασία με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Είχα την ευκαιρία να συναντήσω τον κύριο Γκούσταυσον και τον κύριο Ταραμπέλα στην επίσκεψή σας το Νοέμβριο πέρυσι στην Κοπεχάγη και ύστερα από την ε, επικοδομητική μας συνάντηση με χαρά έρχομαι να σας παρουσιάσω την, ε, το πρόγραμμα της προτάσεις για ε, την ισότητα μεταξύ των φίλων. Συμβούλιο έχει επιλέξει ε, τα συνθήματα υπεύθυνη Ευρώπη, ισότιμη Ευρώπη, πράσινη Ευρώπη, δίκαιη Ευρώπη, που βέβαια καλύπτει και την ισότιμη μεταχείριση και τα δικαιώματα των γυναικών. Πρόκειται για συνθήματα Ε, δίνουν βέβαια τις προθέσεις της ε, Προεδρίας ε, της Δανίας και το πρόγραμμα για την ισότητα των φίλων έχει να κάνει με οικονομική αλλά και κοινωνική πολιτική. Για να προχωρήσουμε με έναν τρόπο δυναμικό, πράσινο και υπεύθυνο θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερο ρόλο και στην ε, ισότιμη μεταχείριση των φύλων. Η ισότητα των φύλων είναι βασική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να καθησυχάσω, να διαβεβαιώσω την Επιτροπή σου θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για να εξασφαλίσουμε πρόοδο και να συμβάλλουμε στις σημαντικές ε, στο μέγιστο δυνατό βαθμό ε, στο σημαντικό αυτό θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίω έχουμε προχωρήσει πολύ, αλλά ακόμη πολλά μένουν να γίνουν και σε αυτέ τι εποχέ τη κρίση. Η μεταχείριση ανδρών και γυναικών έχει τεράστια σημασία. Πρέπει να αξιοποιήσουμε κάθε ικανότητα, τάλαντο, ε, δεξιότητα από το εργατικό μα δυναμικό. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια μόνο οικονομία, σημαίνει ταυτόχρονα και ανθρώπινα δικαιώματα, σημαίνει ταυτόχρονα και ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Δεν μπορούμε να μεταχειριζόμαστε του ανθρώπου διαφορετικά μόνο και μόνο ε, λόγω του φίλου τους. Πρέπει αντιθέτω ε, να βεβαιωνόμαστε πάντοτε ότι κάθε πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα έχουν ίσα δικαιώματα και στις ευκαιρίες. Κανεί δεν μπορεί να υφίσταται διακρίσει λόγω του φίλου του. Κυρίε και κύριοι τη Επιτροπή, η βία κατά των γυναικών είναι ένα από τα κύρια προβλήματα που εμφανίζονται σε όλε τι χώρε, σε όλε τι περιοχέ του κόσμου και σε όλα τα στρώματα τη κοινωνία. Πρέπει λοιπόν να διαρρήξουμε τα ταμπού, να καταστήσουμε σαφές ότι δεν είναι αποδεκτή η βία. Αντιβαίνει όχι μόνο στον νόμο, αποτελεί σοβαρή ζημιά, προξενεί σοβαρή ζημιά στο άτομο, στον πολίτη, στην προσωπικότητά του. Είναι ένα ζήτημα το οποίο γνωρίζω ότι ενδιαφέρει ιδιαίτερα κάποιους από τους βουλευτές της Επιτροπής σας και θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω, καθώς έχω εργαστεί ως κοινωνικός λειτουργός τα τελευταία 20 χρόνια ε, στη σταδιοδρομία μου, το θέμα της ε, βίας κατά των γυναικών, ε, της ενδοοικογενειακής βίας, είναι θέμα που έχω, για το οποίο έχω, στο οποίο έχω ιδιαίτερα αφοσιωθεί. Πρέπει οι γυναίκες να αισθάνονται ασφάλειες στα σπίτια τους και τα παιδιά δεν πρέπει να εκτίθενται στη βία που προξενεί πολλά προβλήματα στην υγεία τους. Πρέπει λοιπόν να υπενθυμίσουμε ότι δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Έχουμε πρωτοβουλίες που ήδη έχουν ξεκινήσει, έχουν εκτελεστεί, έχουν εξασφαλιστεί σημαντικές πρόοδοι. Φερρυπίν, πέρυσι η Επιτροπή με μια μελέτη του Ευρωβαρόμετρου για την ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών διαπίστωσε ότι 9% 90% των πολιτών τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν υψηλό βαθμό επαγρύπνηση και ευαισθητοποίηση ω προ την ενδοοικογενειακή βία εις βάρος των γυναικών. Αυτό σηματοδοτεί μια πολύ σημαντική αλλαγή συμπεριφοράς, νοοτροπία, που είναι προπόθεση για την καταπολέμηση του προβλήματο. Ξέρω επίση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αφοσιωμένη στο στόχο τη ανάπτυξη μια αποτελεσματική πολιτική για την καταπολέμηση τη βία κατά των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ιδιαίτερα καταγράφεται στο πρόγραμμα δράσεων που εφαρμόζεται μέσα από το πρόγραμμα τη Στοκχόλμη για τις γυναίκες, τα παιδιά και την ε, ισότιμη μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών 2010-2015. Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφωνούν ω προ την ανάγκη να καταπολεμηθεί η βία ει βάρο των γυναικών. Η πρόληψη, υποστήριξη προ τα θύματα, αλλά και ε, σκληρές ποινές, ε, κυρώσεις αποτελούν ένα σύνολο για μια κοινή προσέγγιση. Πρέπει και στους τρει τομεί να προχωρήσουμε για να αποδώσουμε τους απαιτούμενους για την πρόοδο πόρους. Κυρίε και κύριοι, κατά τη δανεική προεδρία στο Συμβουλίο θα επικεντρωθούμε σε τέσσερα βασικά κεφάλαια, τα οποία θα επιδιώκουμε πρόοδο και είναι η υποεκπροσώπηση στα διοικητικά συμβούλια των ε, εταιριών γυναίκες, ε, των γυναικών, το, η κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον, ε, η συμμετοχή των γυναικών βέβαια στα προβλήματα αυτά, η διάσκεψη της ε, Νέας Υόρκης και θα ήθελα κυρίες και κύριοι να επανέλθω στο πρώτο θέμα για να αναφερθώ στην ανάγκη να εξασφαλιστεί μια ισότητα μεταχείριση των, ε, αντιμετώπιση και συμμετοχή των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια. Μόνο 60% των πτυχιούχων Ε, πανεπιστημίων ε, ήταν ε, γυναίκες. Το 45% της κοινωνίας είναι γυναίκες και η συμμετοχή των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια αποδεικνύει ότι είναι πάρα πολύ χαμηλή. Χρειάζεται μια καλύτερη λοιπόν εξισορρόπηση μεταξύ των φύλων όσον αφορά την λήψη υπόψη των δεξιοτήτων και προσόντων κατά την ανάθεση μιας θέσης εργασίας. Η παρουσία των γυναικών ε, σε διοικητικά συμβούλια εταιριών αποδεδειγμένα βελτιώνει τις επιδόσεις ε, μιας επιχείρησης και γι' αυτό η Δανία ε, θέλει να αναλάβει δραστήρια συμμετοχή το Συμβούλιο στο θέμα αυτό, στη συζήτηση του θέματος αυτού σε διάσκεψη που θα γίνει σύντομα και σκοπεύουμε να συζητήσουμε λύσεις και προτάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Η Δανία η Δενική Προεδρία θέλει να στηριχθεί στην ευέλτιστη εμπειρία των κρατών και να επιτρέψει το Συμβούλιο να συζητήσει το τι μπορεί να γίνει για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της υποπροσώπησης και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών. Επίσης, το Συμβούλιο έψω θα ε, καταθέσει τι προτάσει του ω προ την αυτορύθμιση και τι προτάσει για τη του ζητήματο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ξεκινήσει η συζήτηση το Μάρτιο. Η Δανία, η Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο θα υποδεχθούν από κοινού μια ανταλλαγή ευέλθυνων πρακτικών ε, για τι γυναίκε στη λήψη των αποφάσεων, μια, μια εκδήλωση που θα γίνει εφέτο στο Όσλο τη Νορβηγία. Επίσης, κατά τη διάρκεια της Δανικής Προεδρίας ε, θα αναπτυχθεί και η παρακολούθηση των, ε, της συνέχισης της ε, πλατφόρμας του Πεκίνου για δράση που θα επικεντρωθεί σε ένα γεγονός που δεν έχει αντιμετωπιστεί ακόμη, το περιβάλλον δηλαδή, η σχέση της γυναίκας με το περιβάλλον, το τομέα ΣΚΑΠΑ. Και έτσι στη ισότιμη μεταχείριση και την κλιματική αλλαγή πάλι θα υποβληθεί το θέμα αυτό στο Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ ε, τον Ιούνιο. Επίσης, νέους δείκτες. Νέους δείκτες που θα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ήθελα να σημειώσω ότι με χαρά διάβασα την έκθεση της κυρίας Κιλνίλσον για τις γυναίκες και την κλιματική αλλαγή. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Οι γυναίκες και οι άνδρες δεν έχουν ισότιμη μεταχείριση στη λήψη των αποφάσεων σε θέματα σχετικά με τις κλιματικές αλλαγές. συμπεράσματα του Συμβουλίου περιλαμβάνουν δείκτες που δεν αναμένεται να, που αναμένεται να επικεντρώνεται σε δύο πράγματα. Η συμμετοχή ε, των γυναικών στην ε, μηχανολογική ε, σχεδιασμό πόλεων, μαθηματικά, φυσικομαθηματικά και τη σχέση με την κλιματική αλλαγή. Ο τρίτο τομέα είναι η κατάρτιση και η εκπαίδευση των γυναικών. Μεγάλη πρόκληση για αρκετέ χώρε. Πολλέ ε, κοπέλε αλλά και αγόρια δεν μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα με βάση τα προσόντα του και τα ενδιαφέροντά του το χώρο στον οποίο θα σπουδάσουν. Είναι υποχρεωμένα να ακολουθήσουν δηλαδή τις ε, παγιωμένες προσδοκίες σε σχέση με το κάθε φύλλο. Η Ιδανική Προεδρία λοιπόν προσπαθεί να εξετάσει και το θέμα αυτό και υπό τη αυτή να αναζητήσει λόγους του οποίους κάποια νέα παιδιά εγκαταλείπουν το σχολείο με την ετήσια διάσκεψη της, ε, με την ετήσια συνάντηση της διάσκεψης για τα δικαιώματα των γυναικών θα συζητήσουμε και την χειραφέτηση των γυναικών, την πρόσδοση εξουσίας στις γυναίκες αλλά και την απαλλαγή τους από τη φτώχεια και την εξαθλίωση. Έτσι λοιπόν μαζί με την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ιδανική Προεδρία θα προσπαθήσει να εξασφαλίσει πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, στις, ε, στα συμπεράσματα αλλά και στα ψηφίσματα τα ε, αγαπητά μέλη της, Ευρωπαϊκής, της Επιτροπής σας, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ παρόντες και που μου δίνετε την ευκαιρία να σας μιλήσω σήμερα. Πριν όμως περάσω στη συζήτηση, θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Φάιξεν, ε, συνάδελφο Υπουργό για θέματα απασχόλησης. Ευχαριστώ θερμά. I Ξεκινώντας, ε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση Είμαι ευτυχής που βρίσκομαι ανάμεσά σας ε, και ελπίζω πως θα έχουμε μια ανοιχτή και ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων για τους επόμενους έξι μήνες. Η Ιδανική Προεδρία του Συμβουλίου φτάνει σε μια πολύ σημαντική στιγμή τόσο για την Ευρώπη όσο για το υπόλοιπο κόσμο. Η κρίση έχει πλήξει σκληρά την Ευρώπη και δυστυχώς θα συνεχίσει θα υπάρξουν πολλές επιπτώσεις ε, για χιλιάδες άνδρες και γυναίκες ε, που χάνουν ή φοβούνται ότι θα χάσουν την θέση τους στην εργασία. Μόλις είπε ο συνάδελφός μου ότι η ισότητα ανάμεσα στους άνδρες και γυναίκες είναι ένα θεμελιώδες ε, στοιχείο για την κοινή θεμελιώδη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αντίθετα από άλλε περιοχέ του κόσμου, έχει διασφαλίσει την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στον τομέα τη εργασία. Φυσικά, αυτό είναι σημαντικό, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε πω πολλά απομένουν να γίνουν ακόμα. Ω Υπουργό Απασχόληση ε, στη Δανία, συχνά ε, αντιμετωπίζω διάφορε περιστάσει ε, ανισότητα δηλαδή, στην Δανία. Μιλάμε για ε, αμοιβέ ε, για προαγωγέ ε, και ούτω καθεξής. Κάθε φορά πρέπει να ε, σας πω ότι εκπλήσωμε ότι πως τον 21ο αιώνα πρέπει να πείσουμε ακόμα τον κόσμο ότι άνθρωποι και γυναίκες έχουν τα αυτά δικαιώματα. Ιδιαίτερα σε εποχές κρίσης δεν πρέπει να αφήσουμε της θεμελιώδη αρχή της ε, ισότιμης αντιμετώπισης και μεταχείρισης να υποβαθμιστεί. Ως υπουργό Απασχόλησης επιθυμώ να υπογραμμίσω την σημασία της γυναικείας συμμετοχής ε, στον αγορά εργασίας. Οι γυναίκες στην αγορά εργασίας ε, συμβάλλουν σημαντικά στην ευημερία της Ευρώπης. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν η στρατηγική 2020 τονίζω, τονίζει τη σημασία ανδρών και γυναικών και την αυξημένη τους συμμετοχή στην αγορά εργασίας. Είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε ότι αν τις γυναίκες ε, συμβάλλουν με τον αυτό τρόπο και ω εκ τούτου πρέπει να έχουν και τα αυτά δικαιώματα. Πρέπει να το έχουμε πάντα κατά νου όταν εξετάζουμε οδήποτε ζήτημα που άπτεται της αγορά εργασία η Δανία θέλει να υποστηρίξει την ευφυή ε, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμό ε, οικονομική ανάπτυξη την ε, και θέλει να ασχοληθεί με το ζήτημα της συνοχής στον τομέα της αγοράς εργασίας. Να αναφερθώ τώρα στην ίση αμοιβή ανδρών γυναικών στην αγορά εργασίας κρίνω πως ε, η αμοιβή είναι μια θεμελιώδης αρχή, γι' αυτό θα πρέπει να εργαστούμε ε, για αυτήν. Άνδρες γυναίκες ε, έχουν τα ίδια δικαιώματα σε ό,τι αφορά την αμοιβή. Αυτό αποτελεί μια πρόκληση θα λέγαμε Γνωρίζω πως ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμεί η Κομισιόν να εξετάσει το ζήτημα της ίσης, της ίσης αμοιβής και το 2012 πρόκειται να υποβάλει μια σύσταση προς την Κομισιόν. Ε, νομίζω ότι αυτή η σύσταση θα είναι ένα πολύ καλό εργαλείο για περαιτέρω δουλειά επί του προβλήματος. προβλήματος. Κατά τη διάρκεια της Δανικής Προεδρίας ε, προγραμματίζουμε μια διάσκεψη τον Μάιο, τον Μάιο σχετικά με πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε περιπτώσεις που παραβιάζεται αυτή η αρχή. Έχει αποδειχθεί σε πολλές περιπτώσεις δύσκολο για τους ε, ανθρώπους που έχουν υποστεί διακριτική μεταχείριση να την διεκδικήσουν ε, σε επίπεδο εργοδοσίας. Η διάσκεψη του Μαΐου θα έχει ως στόχο αυτό ακριβώς ε, το στοιχείο και ελπίζω πολλοί από εσά να μπορέσουν να συμμετάσχουν. Μια, μια ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική ζωή και τον ιδιωτική ζωή, την προσωπική ζωή, είναι κάτι το οποίο ανέκαθεν ζητούσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πολύ καλές πρωτοβουλίε ε, έχουν αναλυφθεί, ε, άδειε μητρότητας, και από αυτό έχουν οργανωθεί και πολλέ διασκέψει. Ένα άλλο ζήτημα που θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι οι δύο γονεί χρειάζεται να έχουν ευκαιρία να παίρνουν γονική άδεια ενώ τα παιδιά τους είναι ακόμα νέα, μικρά. Και αυτό για το καλό των παιδιών και των οικογενειών, αλλά και για μια καλύτερη εκπληκτική ισορροπία ανάμεσα στους άντρες και γυναίκε. γυναίκες. Και τέλος, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, δεν χρειάζεται να επενθυμίσω στην Επιτροπή ότι το σχέδιο οδηγίας για την άδεια μητρότητος δεν είχε μια εύκολη ζωή. Οι συζητήσεις στο Συμβούλιο μερικές φορές ήταν ιδιαίτερα τεταμένες και όλοι γνωρίζουμε εδώ σήμερα ότι οι τροπολογίες που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Οκτώβριο του 2010 δεν κατέθεσαν ε, την ζωή αυτής οδηγίας ευκολότερη και οι τροπολογίες ε, για την ε, θέμα της ε, ίσης αμοιβή δεν ήταν κάτι το οποίο μπόρεσε ευκόλως να αποδεχθεί το Συμβούλιο. Όπως γνωρίζετε υπάρχει μια μειοψηφία η οποία μπλοκάρει τις περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Ως Προεδρία θεωρούμε ότι η σημερινή κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς συμφωνείτε αλλά επίσης ε, θεωρούμε ότι είναι δυστυχές το γεγονός διότι δεν συμβάλλει σε μεγαλύτερη συνεργασία ανάμεσα στο Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Ως Προεδρία θα ήθελα να διερευνήσω αν υπάρχουν δυνατότητες για έναν ε, περαιτέρω διάλογο επί του θέματος. Ταυτόχρονα θα πρέπει να επενθυμίσω τις δυσκολίες που το Συμβούλιο αντιμετωπίζει και εγώ πρέπει φυσικά να σεβαστώ τις ε, ιδέες οι οποίες προέκυψαν από το τελευταίο Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ το 2011. Η έκθεση προόδου αναφέρει ότι θα πρέπει να υπάρχουν περαιτέρω διαβουλεύσεις με την Κομισιόν και το Ευρωκοινοβούλιο ως ε, ένας τρόπος προκειμένου να αναζωογονηθεί ο διάλογος μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Γι' αυτό λοιπόν ελπίζω ως ε, αρμόδια υπουργό το Ευρωκοινοβούλιο να συμμετάσχει σε έναν επικοδομητικό διάλογο με την Προεδρία αναφορικά με το πώς θα σπάσουμε τον πάγο. Αυτό θα είναι ένα από τα έργα που θα αναλάβω αυτές κατά διάρκεια της Προεδρίας μου και ελπίζω να επιτύχουμε την επιθυμητή πρόοδο. Θα πρέπει να τονίσω επίση και τη σημασία που αποδίδει το Συμβούλιο στην ανάγκη για μεγαλύτερη ευελιξία και συμβαστικό πνεύμα από πλευρά Ευρωκοινοβουλίου, εάν οι άτυπε διαπραγματεύσει στεφθούν υπό επιτυχία. Αυτά είχα να πω ω εισαγωγή. Ελπίζω πως η σημερινή συζήτηση θα έχει μια επικοδομητική ανταλλαγή απόψεων επί των ζητημάτων που έφυξα αλλά και επί των φακέλων που εκκρεμούν και οι οποίοι χρήζουν περαιτέρω εργασία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε πώς βλέπετε εσείς τα πράγματα mm-hmm. και αναφερθήκατε σε πολύ σημαντικά θέματα στα οποία εργάζεται η Επιτροπή μας και στα οποία προσπαθούμε να προχωρήσουμε. Έχουμε τώρα ένα μακρύ κατάλογο ρητών. Ίσως στην αρχή δεν ήμουν αρκετά σαφής. Πάντως ε, ήθελα να πω ότι πρώτα θα δώσουμε το λόγο συντονιστές και μετά στα άλλα μέλη της Επιτροπής. Και υπάρχει μια πρόταση να έχουμε περιορισμένο χρόνο αλλά έχουμε αρκετό χρόνο μπροστά μα. Εάν λοιπόν δεν υπερβάλλετε και προσπαθείτε να λάβετε υπόψη και άλλοι θα θέλουν να μιλήσουν, θα μπορούμε να είμαστε νομίζω ευέλικτη. Αλλά ας μην με μακρηγορήσουμε. 20 έχω εγγραμμένο στο κατάλογο των αγορητών. Και... Ε, ε, Καταρχήν συντονιστέ έχουν το λόγο λοιπόν. Η κυρία Νελεσίβα. Αλλά πρώτα η κυρία Τόμψον από του σοσιαλιστές. Δεν ξέρω τι να μιλήσω. Αγγλικά, δανέζικα, ό,τι προτιμάτε. Α, αγγλικά τότε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε εδώ στην Επιτροπή μας. Είμαστε πολύ ευτυχείς που έχουμε την ευκαιρία να έχουμε ένα διάλογο μαζί σας πάνω στα τόσο σημαντικά θέματα που θίξατε στις ε, τόσο ενδιαφέρουσες εισαγωγικές σας παρατηρήσεις. Θα ήθελα να συγκεντρώσω την προσοχή μου στην άμυση, άνηση συγγνώμη, αμοιβή γιατί αυτό είναι ένα πολύ καυτό θέμα του επόμενου μήνε στην Επιτροπή μα. Ξέρουμε ότι η μη ίση αμοιβή οφείλεται σε διάφορου παράγοντε στα διάφορα κράτη-μέλη. Ίσως λόγω τη δομή τη αγορά απασχόληση. πρότυπα ίσω ε, στην, ε, σε μια χώρα που στην Πορτογαλία έχουν μόνο 8% διαφορά. Σε άλλες χώρες είναι 30%. Στη Δανία, παραδείγματος χάνει 17% είναι η διαφορά αυτά της πληρωμής ανδρών και γυναικών. Ξέρω βέβαια ότι και οι δύο ενδιαφερόσαστε. Και ένα πάρα πολύ σημαντικό παράγοντα είναι ότι η αγορά απασχόληση είναι χωρισμένη ανάλογα με το φύλλο. Και έχουμε τώρα μια νέα ευκαιρία στην Ευρώπη. Γιατί όπως είπε ο υπουργό για την ισότητα όταν αναφέρθηκε στις γυναίκες και το περιβάλλον, στις γυναίκες και τις κλιματικές αλλαγές, στην ανάγκη να συμμετάσχουν οι γυναίκες στην αναπτυσσόμενο κόσμο. Ναι, όλα αυτά τα υποστηρίζουμε. Αυτό που μας φαίνεται όμως πολύ ενδιαφέροντα, έρχομαι μόλις από μια συνάντηση που είμαι η συγγήτρια της... Ε, ε ομάδας μου για την ε, οδηγία για την αποτελεσματική χρήση ενέργεια. Η Κομισιόν λέει ότι θα δημιουργηθούν 2 εκατομμύρια νέε θέσει απασχόληση και ξέρουμε ότι στον τομέα τη ενέργεια το 80% των θέσεων απασχόληση είναι αρσενικέ θέσει, αν θέλετε, που τι έχουν άντρε. Και δεν μπορούμε τώρα να δεχθούμε 2 εκατομμύρια νέε θέσει απασχόληση, εκ των οποίων το 80% θα πάει σε άντρε. Με την κρίση που έχουμε στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, έχουμε εδώ μία τεράστια ευκαιρία να ε, καταρρύψουμε αυτή την διάκριση στην αγορά απασχόληση στην Ευρώπη. Αυτό πρέπει νομίζω να είναι μια προτεραιότητα της ε, ε, Προεδρίας. Στις 27 Φεβρουαρίου εδώ στην Επιτροπή μας θα έχουμε μια διάσκεψη για τις γυναίκες και τις πράσινες θέσεις εργασίας. Πώς θα μπορούμε δηλαδή να περάσουν έτσι οι γυναίκες στον ε, τομέα ανάπτυξης και να μην είναι εκείνες που θα χάσουν από την κρίση. Η δημιουργία θέσεων απασχόλησης θα πρέπει να έχει και μία διάσταση φύλου. Γιατί πολλές φορές ο τύπος των θέσεων εργασίας που συζητάμε είναι ανδρικές εργασίες, ε, ε, θέσεις εργασίας και δεν συζητάμε πώς θα μπορούν να ε, εποφιλθούν οι γυναίκες. Λοιπόν, αυτός είναι ένας από τους πολύ σημαντικούς το παράγοντες της άνησης ε, μεταχείρισης, νομίζω. Ευχαριστώ. Πρώτα σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τρία λεπτά μιλήσατε. Πολύ ωραία. Αν και οι 20 μιλήσουν από τρία λεπτά, μια ώρα δηλαδή, θα είμαστε πολύ καλά. Η κυρία Μπρόνα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστώ τους διευπουργούς που ήρθαν εδώ για να μας αποθύνουν το λόγο. Χάρηκα που άκουσα ε, αυτά που έχει να μας πει ο κύριος Σαρίν. Ε, πραγματικά έχετε πολύ παλιό ιστορικό για την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών. Ως εισηγήτρια για το θέματα των θυμάτων. Είχα την ευκαιρία να συναντήσω την Δανική Προεδρία και εκπροσώπους επίσης του Δανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ο κύριος Πόσκοφ, αν ε, προφέρω σωστά το όνομά του, υπουργό Δικαιοσύνης, είδα ότι είναι πάρα πολύ ε, πρόθυμος να δεσμευτεί εδώ. Βέβαια, ξέρουμε ότι η πρόταση του Συμβουλίου είναι πολύ ε, περιοριστικό. Όχι μόνο αποκλείει τη βία βάση του φύλου από τη δέσμη αυτή, αλλά και σε άλλα θέματα είναι πολύ περιοριστικό όσον αφορά την ενημέρωση, κάποια βασικά δικαιώματα των θυμάτων, παραδείγματο χάρη. Πώς σκοπεύετε να προσπίσετε δική μας θέση. Δεν υπήρχε τίποτα το πολύ εύκολο εδώ όσον αφορά τις προτεραιότητες που δίνει η δική μας Επιτροπή. Κυρία Φρεντερίξεν, είπατε ότι είναι δύσκολο το θέμα της άδειας μητρότητα, μα όλα είναι δύσκολα. Κάθε βασική προτεραιότητα που δίνουμε εμείς στην Επιτροπή μας είναι προβληματικό θέμα για το Συμβούλιο. Πώς σκοπεύετε λοιπόν να αντιμετωπίσετε θέματα που ζητούν οι Ευρωπαίοι πολίτες από εμάς και θα πρέπει πραγματικά να τους τα δώσουμε. Άσχετα από ποια είναι η θέση κάθε φορά του Συμβουλίου, εμείς πρέπει να δώσουμε αυτά τα αποτελέσματα. Τι σκοπεύετε λοιπόν να κάνετε γιατί σήμερα συνάντησα τον εισηγητή στην Επιτροπή Τζούρι και οι εισηγητές της Τζούρι, της Λίμπη και της ΦΑΜ. Και είμαστε πρόθυμοι να προστατεύσουμε τα θύματα της βίας που βασίζεται στο φύλλο, αλλά θα πρέπει να δούμε πώς θα προχωρήσουμε έναντι του Συμβουλίου. Υπάρχει πολλή πίεση από ομάδες πίεσεων. Τι σκοπεύετε να κάνετε εσείς, έχετε κάποιο πρόγραμμα. Θέλουμε όμως να ολοκληρώσουμε η διαδικασία της πρώτης ανάγνωσης κατά διάρκεια δικής σας προεδρίας. Φιλόδοξο μεν, αλλά νομίζω θα πρέπει να το κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρος. Η κυρία κορνέλη έχει το λόγο. Προσπαθώ να συνοψίσω για να αφήσω χρόνο και τους συναδέλφους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μια από τις προκλήσεις προεδρία θα είναι η διαπραγματεύσει στο ΕΠΣΚΟ και στο Εαρινό Συμβούλιο για τι προτεραιότητε για την αληθινή ε, οικονομία, την αγορά εργασία το 2012, το δεύτερο εξάμεινο. Και ναι, μεν, ε, πρόκειται για θέματα που έχουμε επεξεργαστεί. Εύρετα όμω επικρατεί η αίσθηση ότι οι οικονομικές ανησυχίες τείνουν να επικρατούν των κοινωνικών και λοιπόν ανησυχιών. Θα έλεγα λοιπόν ότι εσείς, η Δανική Προεδρία, ίσως και η Σουηδική και κάποιες ώρες ε, και άλλες χώρες που ε, αντιλαμβάνονται ποια είναι η κατάσταση. Φερρυπίν ότι δεν έχει δίκιο η Γερμανία με τη μονομανία της, για να είμαστε ειλικρινείς, ότι μόνο η δημοσιονομική εξυγίανση μπορεί να δώσει τη λύση. Η μου η Ευρώπη μπορεί να θεωρούν οι Γερμανοί ότι αποτελείται από επιχειρήσει, αλλά η δικιά μου αποαρτίζεται από ανθρώπους και από αυτούς οι μισοί είναι γυναίκες. Ελπίζω λοιπόν ότι η Προεδρία της Δανίας θα είναι στο πλευρό μας στην υπόθεση αυτή και θα ήθελα η έκθεση που θα ε, εγκρίνει το Κοινοβούλιο και τις οποίες τιμή έχω εγώ να, να αναλάβω την σύνταξη έχω εγώ τιμή να έχω την ε, σύνταξη θα ε, σας στηρίξει στις προσπάθειές σας και για τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, του Ερενού Συμβουλίου για την προστασία των παιδιών την ε, μέρημνα για τα παιδιά ιδιαίτερα, δηλαδή ε, τη δυνατότητα που, γίνεται, που δίνεται στη γυναίκα να εργάζεται εφόσον παρέχεται επαρκή φροντίδα και μέρημνα για τα παιδιά. Γιατί οι προτάσει για περικοπή των σχετικών δαπανών δεν βοηθάνε καθόλου στην παραμονή τη γυναίκα στον χώρο εργασία. Πιστεύω ότι πολλά πράγματα θα έπρεπε να έχουν γίνει και δεν έχουν γίνει ακόμη αρκετά και ελπίζω ότι θα μπορέσετε να πιέσετε και σε από πλευρά σας μια ακόμη συνάντηση μέσα στο εξάμεινο που θα υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι το θέμα αυτό για άλλη μια φορά. Δεν νομίζω ότι θα μας βοηθήσει. Πιστεύω ότι ό,τι νομοθεσία έχει θεσπιστεί πρέπει να υλοποιηθεί ουσιαστικά.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 τον επιχειρηματικό κλάδο και για κάποιον που πρόκειται από τον κλάδο αυτό θεωρεί τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ως ε, τον τρόπο προκειμένου να προχωρήσει η επιχειρηματικότητα των γυναικών και αν ε, έχετε κάτι υπόψη σας αναφορικά με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πώς μπορούμε να προωθήσουμε τη συμμετοχή των γυναικών στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ένας άλλος κλάδος που με ενδιαφέρει είναι η ε, αναφορά που κάνετε στις, ε, στα ποσοστά. Εγώ είμαι κατά των ποσοστών, εγώ θέλω περισσότερες γυναίκες φυσικά στα διοικητικά συμβούλια, αλλά θεωρώ πως το δανέζικο παράδειγμα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Και ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο είναι το ότι στη Δανία ασχολείται με την διαφορετικότητα, την ετερότητα. Και δεν μιλάμε μόνο για τις γυναίκες, αλλά και τι εθνικές μειονότητες, διάφορες εθνότητες κλπ. Θα μπορούσατε να μας πείτε κάτι παραπάνω. Ευχαριστώ. Κύριε ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ε, ερώτηση που θέλω να κάνω αφορά την ε, αναγκαιότητα σχετικά με την καταπολέμηση και της κρίσης. Κρίση η οποία πλήττει ιδιαίτερα έντονα την χώρα μου, την Πορτογαλία και αυτό φυσικά όπως καταλαβαίνετε πλήττει και το δικαίωμα στην εργασία και τα κοινωνικά δικαιώματα κάτι το οποίο επηρεάζει άμεσα και τα δικαιώματα των γυναικών. Αυτή είναι μια από τις ανησυχίες για όλους όσοι υποστηρίζουν τα δικαιώματα των γυναικών. το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η κυβέρνηση της Πορτογαλίας συμφώνησαν επί μέτρων τα οποία θα διευκολύνουν τις απολύσεις και όπως αντιλαμβάνεστε αυτό θα καταστήσει ακόμα πιο επισφαλή τη θέση των γυναικών στην αγορά εργασία και θα οδηγήσει σε μια γενικότερη αύξηση της ανεργίας. Και αυτό άπτεται όπως είναι φυσικό και με τα δικαιώματα των γυναικών, διότι είναι πολύ δύσκολο να υποστηρίξουμε τα δικαιώματα μιας εργαζόμενης όταν η εργαζόμενη αυτή έχει λιγότερες δυνατότητες να υποστηρίξει τη δικαιώματά της και ενδέχεται να δεχθεί κάποιες περικοπές, ε, κάποιους περιορισμούς ε, και στην μητρική άδεια, στην εμπάδια μητρότητας κλπ. Στην Πορτογαλία συμφωνήσαμε, δεδομένη της οικονομικής κρίσης, ε, οι εργαζόμενοι να εργάζονται περισσότερο χρονικό διάστημα ημερησίως, μέχρι 12 ώρες ημερησίως έως και 100 ώρες εβδομαδιαίως. Είναι απαραίτητο λοιπόν να υποστηρίξουμε τα δικαιώματα των γυναικών διότι και αυτές έχουν ε, δικαίωμα συμμετοχής ε, στα κοινά, συμμετοχής ε, στην πολιτική κλπ. Θα ήθελα να γνωρίζω τι πιστεύουν οι υπουργοί πάνω σε όλα αυτά τα ζητήματα η όπως καταλαβαίνετε επηρεάζεται η κατάσταση στα κράτη-μέλη και από τη θέση που κρατούν οι υπουργοί σε άλλες χώρες. Πρώτον να δώσω το λόγο λοιπόν στους ε, επόμενους ε, συναδέλφους. Νομίζω πως ε, θα πρέπει να απαντηθούν, να δούμε όμως πώς θα κανονίσουμε το γύρο των ερωταποκρίσεων η κυρία Νίντερ Σέμπερν που είναι συντονίστρια από το και μετά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Δανική Προεδρία που βρίσκεται σήμερα ανάμεσά μας και που μας παρουσιάζει τις προτεραιότητες και μας δίνει τη δυνατότητα να εμβαθύνουμε επί των ζητημάτων που μας ε, ε, ενδιαφέρουν κατά τη διάρκεια των Ιδανικής Προεδρίας. Θα θίξω κάποια ζητήματα που έθεσαν και οι συνάδελφοί μου, αλλά με κατά τη διαφορετικό τρόπο. Η πρώτη μου ερώτηση αφορά στο γεγονό ότι οι μελέτες κατέδειξαν ότι η κρίση είχε ιδιαίτερα αρνητικέ επιπτώσει στον τομέα όπου οι γυναίκες είχαν υψηλά ποστά. Ε, συμμετοχή ε, στην απασχόληση και άρα την άλλη έχουμε κάποιε μελέτε οι οποίε δείχνουν ότι οι γυναίκε που κατόρθωσαν να διατηρήσουν την ε, θέση του και που έχουν την πλειοψηφία στι επιχειρήσει, αυτέ οι επιχειρήσει μπόρεσαν να αντισταθούν αποτελεσματικότερα στην κρίση. Λοιπόν, η Δανική Προεδρία ενδιαφέρεται στο, με το θέμα αυτό. έχει κάποια ανάλυση που μπορούν, μπορεί να εντοπίσει ποιοι είναι αυτοί οι κλάδοι και να μπορέσουν να καταδείξουν ποιους είναι ο θετικό ρόλο που διαμορφώνουν οι γυναίκε και τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε οι γυναίκε να ξαναβρούν την θέση του, θέση που του ανήκει σε μια ανάπτυξη που θα του είναι ευνοϊκή. Και συμφωνώ εδώ με του συναδέλφου οι οποίοι συνεχάρισαν τη Δανική Προεδρία που έθεσε μεταξύ των προτεραιοτήτων την ισότητα των αμοιβών. Αυτή η πραγματικότητα όμως μας δείχνει ότι άνδρες και γυναίκες για την ίδια εργασία δεν αμείβονται με τον αυτό τρόπο. Και σε ό,τι φορά τώρα την πρωτοβουλία της κυρίας Ρέντινγκ, ειδικά την εκπροσώπηση των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια, η προθεσμία ενό έτου που έδωσε η ίδια η κυρία Ρέντινγκ πέρυσι ε, εκπνέει σε ένα μήνα. Ποια θα είναι η στάση λοιπόν η Ιταλική Προεδρία σχετικά με την εν λόγω πρωτοβουλία που έχει ως στόχο την αύξηση τη συμμετοχή των ε, γυναικών στα διοικητικά συμβούλια και να επιστώ την προσοχή σας επίσης ε, στην καταπολέμηση κατά των στερεοτύπων και των ε, προγραμμάτων ε, εκπαίδευση των νέων κοριτσιών. Ξέρουμε ότι συνήθως τα κορίτσια ασχολούνται περισσότερο με φιλολογικές σπουδές. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε λοιπόν αναφορικά με τις επιλογές τους, διότι είναι ένα ζήτημα το οποίο ε, αφορά και στο νέο δημοσιονομικό πλαίσιο. Έχουμε ένα ερευνητικό πρόγραμμα, θα μπορούσαν να ληφθούν λοιπόν συγκεκριμένα μέτρα και θα μπορούσαμε να στηριχθούμε στην ε, Δανική Προεδρία επ' αυτού. Να επαναλάβω την ερώτηση τώρα σχετικά με την βία κατά των γυναικών και ιδιαίτερα την οικογενειακή βία. Και νομίζω ότι αυτό συνδέεται και με το σωματεμπόριο. Ξέρουμε ότι οι κοπέλες ε, είναι τα θύματα αυτή τη ε, κατάσταση. Θα θέλαμε να γνωρίζουμε ε, στο, εάν στο όνομα τη δανική προεδρία, ε, στο πρόσωπο της δανική Προεδρίας θα έχουμε έναν σύμμαχο για να προχωρήσουμε σε μια πραγματική υποστήριξη αυτών των θυμάτων, διότι βλέπουμε ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο, στο οποίο δεν πρέπει να σταματήσουμε επειδή εγκρίθηκε μια οδηγία ή επειδή εγκρίθηκαν κάποια νομοθετικά κείμενα, κάποια ψηφίσματα. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να συνεχίσει να μας προσχολεί για να φέρουμε μια ουσιαστική λύση. Τώρα, να επιστρέψω την προσοχή σας κάπως εκτός Ευρωπαϊκής Υπήρου, διότι και αυτό εμπίπτει στις αρχές μας, δηλαδή την τομέα της αλληλεγγύης, νομίζω ότι είναι μια από τις βασικές μας αρχές. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε το ρόλο που οι γυναίκες διαδραμάτισαν κατά τη διάρκεια της Αραβικής Άνοιξης και στις προτεραιότητες της δανεική Προεδρίας ε, τονίζεται μια μεγαλύτερη συνέπεια και συνοχή στην πολιτική ανάπτυξη ε, και έναν επαναπροσανατολισμό. Υπάρχουν ε, οικονομικά μέσα τα οποία κατευθύνονται προ την ε, στήριξη των γυναικών και θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή τη Δανική Προεδρία να συνεχίσουν να στηρίζουν τι γυναίκε αυτέ και να μην ξεχνάμε ότι διαδραμάτισαν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο διάρκεια τη επανάσταση και δεν θα πρέπει λοιπόν να χάσουν κάποια πλεονεκτήματα τα οποία έχουν αποκτήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώσαμε την πρώτη, τον πρώτο γύρο ερωτήσεων με τους συντονιστές και θα πρότεινα τώρα να δώσω το λόγο στους δύο υπουργούς για να απαντήσουν. Παρακαλώ. Ποιος θέλει να ξεκινήσει. Ευχαριστώ πολύ. Εξαιρετικές ερωτήσεις σας. Η μεγάλη πρόκληση για μένα τώρα είναι να μιλήσω αργά. Αν τα καταφέρω. Για την πρώτη ερώτηση, κυρία Τόμσον. Την, ε, διακρίσεις ε, μεταξύ ανδρών και γυναικών στον χώρο της υγείας. Συμφωνώ απολύτω. Ε, αυτό είναι και ο λόγο για τον οποίο ε, ζητήσαμε να θεσπίζουμε του δείκτε για την ε, παρουσία ανδρών και γυναικών. Έχετε το δίκιο. Όταν μιλάμε για διάκριση, για διαφορετική μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών, θα πρέπει να αρχίσουμε να τις αντιμετωπίζουμε ήδη από, την, από το επίπεδο των σπουδών. Και αυτό ισχύει για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για ένα γεγονός το οποίο έχουμε συνείδηση, αλλά πρέπει να σημειώσω ότι είναι μία πορεία η οποία δεν είναι μονόδρομη. Η κυρία Τόμσον μίλησε για δουλειές αντρικές. Μα ακριβώς και μόνο το να ε, χρησιμοποιούμε αυτή την ορολογία ενισχύει το πρόβλημα, το επιδεινώνει. Πρέπει δηλαδή να μην υπάρχει χαρακτηρισμό τέτοιο. Πρέπει κάθε άντρα ε, να μπορεί να διαλέξει και γυναικείες δουλειέ. Και να που και εγώ χρησιμοποιώ ορολογία που δεν είναι σωστή πολιτικά. Λοιπόν, σε εκεί έχετε να προσθέσετε κι εσεί κάτι. Για την κυρία Παραβάνοβα. Παβάνοβα. Μιλήσατε για την ε, βία ει των γυναικών. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο ιδιαίτερα με ενδιαφέρει. Η βία είναι απαράδεκτη. Η βία είναι καταδικαστέα και πρέπει να την χάνει ποινική κύρωση κάθε εκδήλωση βία. Σε αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Γι' αυτό πιστεύω ότι ε, μπορούμε να στηριχθούμε στο πενταετές πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο αλλά και η Επιτροπή συμφωνούν στην απόλυτη καταδίκη της βίας βάρος των γυναικών και την προστασία, την παροχή στήριξη στα θύματα. Πρέπει να έχουμε σαφείς διατάξεις στον τομέα αυτών. Και τόσο Επιτροπή όσο και Συμβούλιο έχουν συνεργαστεί πολύ καλά ε, στο θέμα της οδηγίας για την ε, διακίνηση, για το εμπόριο ανθρώπων. Και επίσης την οδηγία που αφορά την προστασία των ανηλίκων. Έχουμε πολύ καλή συνεργασία. Τώρα συνεργάζεται το Συμβούλιο με το Κοινοβούλιο για την διαπραγμάτευση ενός ε, πακέτου μια δυσθέσμης μέτρων που θα ασχοληθεί με την προστασία των θυμάτων και αρμόδιο θα είναι όχι το ΕΠΣΚΟ αλλά το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Ιστορικών. Θα διατυπώσω τις ε, Ανησυχίες μου λοιπόν και στην Επίτροπο Ρέντινγκ, τα έχω καταγράψει άλλωστε και στην ομιλία μου. Και όπως έλεγα, όπως ήδη είπα δημερό σε κάποιους εξημών, πιστεύω ότι ιδιαίτερα σημαντικό είναι να προχωρήσουμε σε μια χαρτογράφηση της κατάστασης, να γνωρίζουμε δηλαδή που εντοπίζεται η βία βάρος των γυναικών, να λέμε ότι είναι απαράδεκτη η βία κατά των γυναικών, ότι δεν διατηθέμαστε ε, να την αποδεχθούμε και πέραν της ορολογίας να δημιουργήσουμε νέες συνθήκες και νέα πραγματικότητα για τα τωρινά αγόρια που θα γίνουν μια μέρα άντρας, να τους ε, ε, κάνουμε να εμπεδώσουν δηλαδή ότι η βία είναι απαράδεκτη. για τη Ρεγκύρια Κορνέλσον και την οικονομική κρίση. Μπα, όχι, δεν μπορώ να διαβάσω τις σημειώσεις μου, μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Όντω είπατε ότι επικεντρωνόμαστε περισσότερο στι οικονομικέ πτυχέ και όχι τόσο στην ισότητα ανδρών και γυναικών, στι κοινωνικέ πτυχέ τη ισότητα ανδρών και γυναικών. Σωστό είναι αυτό και σύμφωνα και με τι προτεραιότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πλην όμω, θα ήθελα να πω ότι όταν μιλούμε για ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και οικονομική διάσταση, Είναι σαν να μιλάμε για δύο διαφορετικά θέματα, όμως οικονομική ανάπτυξη και η ισότητα είναι δύο έννοιες οι οποίες βαίνουν παραλλήλως χέρι-χέρι. Και δεν ε, μπορώ να περιορίσω την έννοια της ισότητας στην απλή περιγραφή δικαιωμάτων. Είναι κάτι το χρήσιμο ισότητα. Δεν την κάνουμε γιατί είναι μια ωραία αρχή, δεν την εφαρμόζουμε γιατί την προβλέπουν οι συνθήκες. Την εφαρμόζουμε διότι είναι μια ιδέα που αποφέρει προς όφελος όλων μας και γι' αυτό συμφωνώ 100% μαζί σας. για την κυρία Γιανακουδάκη. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις Στο θέμα αυτό θα πρέπει να σας ε, παραπέμψω στον συνάδελφο όλα που ασχολείται με το θέμα αυτό. που έχετε στο σχετικό φυλάκιο, αλλά ε, πρέπει να σας πω ότι επεξεργαζόμαστε κατευθυντήριες γραμμές για την ε, προαγωγή του ρόλου των γυναικών ε, σε θέσεις στελεχών, διοικητικών στελεχών των επιχειρήσεων. Τώρα δηλαδή ε, επιχειρήσει που δεν έχουν γυναίκε στα διοικητικά του συμβούλια, στι ανώτερε διευθυντικέ θέσει, στα ανώτερα κλιμάκια, καλούνται να εξηγηθούν, να δώσουν εξηγήσει γιατί. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να έχουμε και μια αντίληψη πραγματικότητα. Οι προόδοι είναι σχετικά βραδίε. Γυναίκε ε, επιχειρήσεων δεν υπάρχουν πολλέ. Αλλά πιστεύω ότι δεν θα ήταν και λίγε οι επιχειρήσει που θα δέχονταν μια γυναίκα γενική Γενικό, Γενικό Διευθυντή. Απλώς είναι βραδεία η αλλαγή νοοτροπίας. Πρέπει να επηρεάσουμε τις νοοτροπίες λοιπόν για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τους στόχους αυτούς. Και ίσως τώρα να δώσω το λόγο στη συνάδελφο. Κοιτάξτε, ο συνάδελφος νομίζω έχει απαντήσει αρκετές ερωτήσεις. Πλην όμως, ε, ως Προεδρία, δεν μπορώ παρά να υπογραμμίσω ότι ιδιαίτερα σημαντικό κρίνουμε τη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση να την αντιμετωπίσουμε, να εξασφαλίσουμε μακροοικονομική σταθερότητα, να διασώσουμε το ευρώ. Και επίσης θέλω να σημειώσω ότι δεν βλέπουμε αντίφαση η ασυμβατότητα μεταξύ της ανάπτυξης ευρωπαϊκής οικονομίας και μιας υπεύθυνη οικονομικής πολιτικής. Αυτό είναι το σημείο κίνησης που ακολουθεί η Προεδρία μας το Συμβούλιο. Αυτή είναι η προσανατολισμή μας ως Προεδρίας. Του τουλεχθέντος αντιλαμβάνομαι ότι και εσείς ως Επιτροπή υπογραμμίζετε πόσο σημαντικό είναι και να αντιμετωπίσουμε τις οικονομικές προκλήσεις, αλλά και να προωθήσουμε τα κοινωνικά δικαιώματα, την ισότητα ανδρών και γυναικών και όπως έλεγα στην αρχή, δεν θεωρώ ότι οι αξίες αυτές είναι αντιφατικές. Θα έλεγα τον αντίον ότι είναι αλληλοσυμπληρούμενες, δεν μπορούμε να έχουμε τη μία χωρίς την άλλη. Και μερικές φορές, ηρωνικά, μπορεί να λέγεται ότι δεν ε, προξενεί δυσκολίε μόνο η οδηγία για τη γονική άδεια. Βεβαίω αντιλαμβάνουμε, όταν μιλάμε για ισότητα ανδρών και γυναικών, Πολλέ ε, φορέ βρίσκουμε προσκόμματα στον δρόμο μας. Μας ρωτάνε αν όντως θέλουμε να προωθήσουμε την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Κοιτάξτε για την ε, ε, Προεδρία είναι μια βασική αξία η προαγωγή των ίσων δικαιωμάτων, των ίσων ευκαιριών. Αποτελεί δε πρόκριμα για την αναπτυσσόμενη ευρωπαϊκή οικονομία, για την ευρωπαϊκή οικονομία. Σε σχέση με κάποιες συγκεκριμένε ερωτήσεις που ετέθησαν για την Πορτογαλία ήδη τη συστήσαμε σήμερα το πρωί. Πρέπει να πω ότι ως εκπρόσωπος της ε, Προεδρίας δεν είμαι βέβαια τι θα μπορούσα να κάνω σε σχέση με απολύσεις στην ε, Πορτογαλία. Αλλά ως Δανή Υπουργό, αν μου επιτρέπετε να μιλήσω για λίγο ως Δανή Υπουργό και μόνο, θα έλεγα ότι αυτό αποτελεί ε, στατικό τμήμα μιας πολύ υπογειογενικής συζήτησης για το κατά πόσον το flexicurity, η ευελίξη ασφάλεια μπορεί να αποτελέσει ε, λύση σε προβλήματα στο χώρο εργασίας. δεν ξέρω πώς μπορεί ο πολίτης να αντιμετωπίζει και να, βλέπει, να κρίνει την πολιτική για την αγορά εργασίας στην Πορτογαλία ή αλλού. Αλλά ε, εγώ ως Δανή μπορώ να πω ότι αν διευκολύνουμε τις ε, κινήσεις απολύσεων, τις απολύσεις από πλευρά των επιχειρήσεων, αν καταστεί πιο εύκολο να απολύει μια επιχείρηση εργαζόμενους, τότε ε, χρειάζεται οπωσδήποτε ένα πολύ πιο γερό δίκτυο ασφαλείας κοινωνικό και επίσης μια εντονότερη εστίαση στην κατάρτιση ώστε να αποκτήσει κανείς περισσότερα προσόντα, δεξιότητες, εφόσον έχει χάσει τις εργασίες του. Και για να ξαναφορέσω, για να ξανα, ε, φορέσω το καπέλο της Δανικής Προεδρίας, θα έλεγα ότι είναι από τα θέματα τα οποία θα, θα ήθελε η Δανική Προεδρία να συζητήσει χωρίς να πιστεύουμε ότι μπορούμε να μέσα σε 5-6 μήνες να αλλάξουμε όλα αυτά τα προβλήματα, την κατάσταση όλα αυτά τα θέματα. Αλλά πάνω απ' όλα όλα αυτά έχουν να κάνουν με τη διαμόρφωση του σχολικού συστήματος, του εκπαιδευτικού συστήματος. Δυστυχώς, όπως είπατε και εσείς δυστυχώς, βρισκόμαστε σε μια δεινή οικονομική κατάσταση. Όμως, Ξέρετε, οι Αμερικανοί λένε never waste a good crisis, ε, να αξιοποιηθείς πάντα μια κρίση όσο μεγάλη και αν είναι. Ε, γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι έχουμε και εμείς να αποκομίσουμε κέρδος από την κρίση αυτή, ιδιαίτερα για τα παιδιά μας, ιδιαίτερα για τους νέους. Θα ασχοληθούμε με τα θέματα αυτά. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα ενσκύψει στην ε, ε, κρίση, θέματα της κρίσης, την εκπαίδευση και την κατάρτιση τη Δευτέρα και οπωσδήποτε πρέπει να δώσουμε έμφαση στους νέους και τα παιδιά αυτή είναι τη, νεολαία που βρίσκεται, που ε, βρίσκεται άνεργη και που μόνο χάρη στην ε, καλύτερη εκπαίδευση και κατάρτιση μπορεί να βρει μια θέση για την αγορά, ε, στην αγορά εργασίας. Ταυτόχρονα με τον τρόπο αυτό μπορούμε να αντιμετωπίζουμε και τις διακρίσεις που επιβάλλονται μεταξύ των φύλων, βελτιώνοντας το επίπεδο κατάρτισης και των γυναικών όπως και των ανδρών. Η πολιτική απασχόληση είναι μια εθνική πολιτική βεβαίως και πρέπει να παραμείνει εθνική. Αλλά καλό θα ήταν ε, στο Συμβούλιο, στο Κοινοβούλιο να ανταλλάσσουμε βέλτιστες πρακτικές, να μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλον εκεί που υπάρχει μια επιτυχία. Για την Προεδρία βασικά αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να ορίσουμε προτεραιότητες και για μας προτεραιότητα είναι μέχρι το 2020 το 75% των ε, πολιτών μας, να, ε, των νέων μας να εργάζεται. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Γιαννάκοβιτς, δεν ξέρω αν... Ε, την κυρία Γιάννα Κουδάκη εννοεί μάλλον ο μιλητής. Δεν ξέρω αν, αναφέρομαι σωστά, αν προφέρω σωστά το όνομά σας, αλλά μιλήστε για τα ποσοστώσεις εσείς. Με συγχωρείτε, είχα λησμονή στην ερώτησή σα. Αλλά συμφωνώ μαζί σα. Καλώ λέει ο πρόεδρο, ε, Νέα ερώτηση. Κύριε Ταραβέλα. Euh, Όπως επενθύμησε και ο Υπουργό κ. Σαρίν, ε, χαίρομαι που μπορώ εδώ στην Επιτροπή Γυναικών μαζί σα να προετοιμάσουμε την ε, ε, Δανική Προεδρία. Συνέντησα την κυρία Φρεντρίξεν και τον κύριο Σαλή και αισθάνθηκα πάρα πολύ τύχη ε, στις επαφές αυτές γιατί είναι σπάνιο να έχει κανένας προοδευτικός ε, υπουργός στη σημερινή Ευρώπη απέναντί του. και θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Κλάς και την κυρία Αντελέτσεβα γιατί βλέπω ότι περιέργως το ΕΛΚ είναι πολύ απόν από τη συνεδρίαση αυτή. Δεν ξέρω γιατί. Αναρωτιέμαι πως υπάρχει κάποια συνάντηση του ΕΛΚ εκτός ε, έδρας. Αλλά βλέπω την κυρία Νέλσεβα, που είναι η νέα συντονίστρια. Πολύ ευχάριστο αυτό. Μπορεί να ξέρετε και αναφέρει η κυρία Φρέντριξεν στο γεγονός ότι υπάρχει ένας πολύ ουσιαστικός ε, φάκελος. Πρόκειται για την άδεια μητρότητα, να μην ξεχνάμε και την άδεια πατρόπιτε. Και έχει δει και ο Υπουργό που λέει ότι στο κοινοβούλιο εδώ υπάρχει μια θέση που ήταν ισχυρή, που είχε πετευχθεί με πλειοψηφία, αλλά υπήρχαν δύο ομάδε. Η μία ήθελε πραγματικά πρόοδο οι άλλοι προσποιόταν ότι για την κρίση δεν μπορούσε να υπάρχει πρόοδος. Πρέπει όμως να υπάρξει πρόεδρος. Και θα πρέπει να, για να προχωρήσουμε να κάνουμε ένας προς τον άλλον από ένα βήμα. Και νομίζω υπό την Ιδανική Προεδρία με ανθρώπους σαν και εσά υπάρχει μια πραγματική ευκαιρία σε, σε πέντε μήνες δεν μα μείνει παρά πέντε μήνες πια μπορούμε να προσεγγίσουμε τις απόψεις λέω ούτως ώστε να υπάρχει μια απόφαση προς αυτό. Αναφέρθηκαν 20 εβδομάδες με, πλήρη, με πλήρες αποδοχές. Ίσως είναι δύσκολο σήμερα αυτό, αλλά θα πρέπει να δούμε, ε, να πούμε ότι για 10 εβδομάδες θα πληρώνεται τουλάχιστον το 80%. Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει 39 εβδομάδες, ε, αλλά λίγες γυναίκες μπορούν να το κάνουν αυτό. Γιατί πέρα από τις πρώτες εβδομάδες δεν ε, πληρώνονται πια επρακώς, άρα δεν μπορούν οι γυναίκες που είναι αδύναμες οικονομικά να πούμε, ας πούμε, τελικά 18 εβδομάδες ε, ε, που θα πληρώνονται σε 80%. Αυτό νομίζω θα ήταν κάτι που θα μπορούσε να πείσει και το Συμβούλιο στην Δανία βρίσκεται σε πέρα από αυτά τα πρότυπα. Προωθείτε τις οικογένειες, τις γυναίκες ε, είναι καλό να αναγνωρίσετε βέβαια και την ε, ε, άδεια πατρότητα, δικαιώματα των πατέρων. Α κάνουμε λοιπόν ένα βήμα ημέν προ για να υπάρξει μια πρόοδο και βασίζομαι πάρα πολύ στην Δανική Προεδρία γι' αυτό. Είμαι σίγουρο ότι μπορούμε να σα έχουμε εμπιστοσύνη. Πρώτα σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ισότεν. Σα ευχαριστώ πρόεδρε. Και ευχαριστώ και του υπουργού για την παρουσίαση τον πρωτερήτο της Ιδανικής Προεδρίας. Θα πρέπει να δούμε πόση σημασία θα ο... δοθεί της Προεδρίας στο θέμα αυτό. ιδίω μια που ξέρουμε ότι θα υπάρχει πρόθεση της αλληλεγγύης μεταξύ των γενών και την ενεργό ε, γέρανση. Οι γυναίκε πολλές φορές ε, τη χάνουν διακρίσεων ει βάρο του ε, στην ε, αγορά εργασία. Γι' αυτό και οι συντάξει των γυναικών είναι χαμηλότερε γιατί εργάζονται σε τομείς που δεν αμείβονται όσο άλλοι τομείς και επίσης αναγκάζονται να σταματήσουν πολλέ φορέ να εργάζονται για να ασχοληθούν με την οικογένειά του. Οπότε πολλές φορές ε, οι γυναίκες αυτές όταν πάρουν σύνταξη ζουν στη φτώχεια. Τι θα κάνει η Δανική Προεδρία για να μειώσει το κενό των συντάξεων μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Εστρέλα παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να αρχίσω ευχαριστώντας ε, τους Δανούς ε, υπουργού και, να τους, και λέγοντάς τους ότι χαιρετίζω τις προτάσεις τους. Ε, οι προτεραιότητες που μας αναπτύξατε είναι πραγματικά ενδιαφέρουσες για όλους εμάς εδώ γιατί είναι σύμφωνες με τα θέματα που συζητάμε. Τη διαφορετική αμοιβή, τα προβλήματα στην αγορά εργασία, την καλύτερη ενσωμάτωση των γυναικών στις, στους τομείς λήψης αποφάσεων των επιχειρήσεων και της πολιτικής. Αυτά είναι θέματα που μας απασχολούν και εμάς και εσάς. Άκουσα αυτό που είπαν οι συνάδελφοι και έχω να πω ότι οι προσδοκίες στην Δανική Προεδρία είναι πάρα πολύ ψηλέ. Ακριβώς σε αυτόν τον τομέα. Εγώ είμαι η συγγήτρια της ε, νέας μορφής οδηγίας για τη λεγόμενη αδιαμητρότητα. Ε, είναι ένα θέμα που με απασχολεί και με ανησυχεί. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστώ την Ελληνική Προεδρία για τη δήλωσή της και ότι ε, δήλωσε ότι προτίθεται να συζητήσει το θέμα αυτό κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας γιατί πρόκειται για ένα φάκελο ο οποίος πραγματικά εδώ και πολύ καιρό εκκρεμεί και το Κοινοβούλιο. Τον Οκτώβριο του 2010 υιοθέτησε ξεκάθαρη θέση με μεγάλη πλειοψηφία. Η θέση αυτή προωθήθηκε στο Συμβούλιο, αλλά δυστυχώς παρόλο στις προσπάθειες των διαφόρων προεδριών και τις δικές μας προσπάθειες βέβαια, δεν προχώρησε το θέμα και θα ήθελα να τονίσω τον θετικό ρόλο της Πολωνικής Προεδρίας η οποία πραγματικά προσπάθησε πάση θυσία να φέρει σε αίσιο πέρας την εξέλιξη του φακελού αυτού. Παρόλα αυτά όμως δεν υπήρξε ποτέ θετική απάντηση από το Συμβούλιο. Είμαστε πράγματι ανοιχτοί, ευέλικτοι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ελπίζει και επιθυμεί να ολοκληρώσει το θέμα το γρηγορότερο δυνατό. Σήμερα ήδη στη συνάντηση των συντονιστών μας αποφασίσαμε να αποστείλουμε μια σχετική επιστολή προς την Ελληνική Προεδρία. για να σας ενημερώσουμε σχετικά να σας ευιστοποιήσουμε, να σας ε, πούμε ξεκάθαρα ότι πραγματικά θέλουμε να υπάρχει μια κοινή θέση για αυτό το θέμα. Παρακαλώ μεταβιβάστε αυτά που σας λέω στο Συμβούλιο. Γιατί πραγματικά θα πρέπει να δώσουμε μια απάντηση στους πολίτες. Γιατί κανένας δεν το καταλαβαίνει γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Βέβαια βρισκόμαστε σε περίοδο κρίσης η οποία δεν διευκολύνει τίποτα. Από την άλλη μεριά δεν επιτρέπεται η κρίση αυτή να χρησιμοποιείται σαν άλοθη για να μην λαμβάνετε καμία απόφαση. Θα ήθελα πραγματικά να πω ξεκάθαρα ότι στην Ευρώπη η πολιτική λιτότητα θα πρέπει να συνοδεύεται από πολιτική αλληλεγγύης θα πρέπει να εξετάσουμε τις ε, δημοσιονομικές επιπτώσεις. Ε. Εάν υπήρχε 1% περισσότερες γυναίκες στην αγορά απασχόλησης, το κόστος των προτάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα καλύπτει το πλήρως. Λοιπόν, η κρίση δεν πρέπει πάντα να είναι ένα άλοθη και να μην παίρνουμε γι' αυτό θετικές αποφάσεις το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Κομισιόν, το Συμβούλιο έχουν υιοθετήσει στρατηγική 2020. Ένας πολύ φιλόδοξος στόχος. Αλλά ένας στόχος που θα μπορούσε να αυξήσει τουλάχιστον κατά 5% τον αριθμό των γυναικών που συμμετέχουν στην αγορά εργασίας. Δύσκολο βέβαια, δεν λέω. Υπήρξε κάποιο πρόεδρος όμως. 16 νομίζω κράτη-μέλη έχουν εκφράσει τη βούλησή του συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ηνωμένο Βασίλειο βάζει τα περισσότερα εμπόδια. Και στη χώρα αυτή υπάρχει τώρα μια δημοσκόπηση όσον αφορά και την εθνική νομοθεσία πάνω στον τομέα. Νομίζω ότι υπάρχουν τώρα προποθέσει για να βρούμε από κοινού μια ικανοποιητική λύση. Θέλουμε πραγματικά να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό κατά τη διάρκεια της Δανικής Προεδρίας. Δεν είναι πολλής χρόνος βέβαια οι έξι μήνες, αλλά θα πρέπει να καλύψουμε την καθυστέρηση που έχουμε και να εκμεταλλευτούμε το χρόνο που έχουμε ακόμα μέχρι το τέλος της Δανικής Προεδρίας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Κυρία Νίτσεν, ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως ε, και ο συνάδελφος Ταραμπέλα, να πω ότι μας ικανοποιεί να αισθανόμαστε με αυτή την πνοή που διαπερνά την Ευρώπη και αφορά τις γυναίκες και τα θέματα περιβάλλοντος. Ε, πάντως, ως εισηγήτρια σχετικά με το θέμα γυναίκες και κλιματική αλλαγή, να πω ότι η έκθεση την οποία έχω συντάξει δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί διότι κάποιες τροπολογίες θα την βελτιώσουν. Σχεδόν όλες οι τροπολογίες που κατατέθησαν δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να εμπλουτίζουν την έκθεση αυτή και από ό,τι φαίνεται θα υπάρξει συνένεση που και αυτό είναι θετικό στοιχείο. Ε, βλέπω στο πρόγραμμα προ Προεδρίας ε, την ε, βούληση για προώθηση των γυναικών στο τομείς της επιστήμης και στους κλάδους της πράσινης οικονομίας, καθώς επίσης και η πρόθεσή σας να βελτιώσει τους δείκτες σύμφωνα με την πλατφόρμα του Πεκίνου. Σε ό,τι αφορά την θέμα της προβληματικής ε, του φύλου στις ενεργειακές μας πολιτικές, ε, πολιτικές μεταφορών και τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής εν γέννη. Ε, υπάρχει έλλειψη στοιχείων, δεδομένων και έρευνας που μας επιτρέπει να λάβουμε υπόψη αυτή τη διάσταση. Και σε ρωτώ, η Ιδανική Προεδρία θα ήταν υπέρ της ε, κατά της μελέτης σχετικά με το συνδέσμους ανάμεσα στην πολιτική μετριασμού του κλίματος και του φύλου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να λάβουμε υπόψη καλύτερα αυτήν τη διάσταση στις μελλοντικέ κλιματικές πολιτικές της Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Παπαδοπούλου. Thank you, Mr. I also Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να καλωσορίσω τους ε, δύο υπουργούς. Συμφωνώ απόλυτα με τις θέσεις τους. Το πρόβλημα είναι ότι ζούμε σε μια οικονομική κρίση και αυτή η κρίση πλήττει τις γυναίκες στον τομέα της απασχόλησης ε, και δημιουργεί πολλά προβλήματα σε ό,τι φορά τη χρηματοδότηση προγραμμάτων όπως το πρόγραμμα Δάφνη αλλά όντας εισηγητρία για το πρόγραμμα 2013 σχετικά με την ηθαγένεια γνωρίζω ότι ένα εκατομμύριο μόνο θα ε, δοθεί για το ζήτημα αυτό και την ευαισθητοποίηση και ρωτώ πώς ε, η ιδανική προεδρία μπορεί να πείσει την Κομισιόν να καταπολεμήσει αυτές ε, τις ασυνέπειες διότι η Κομισιόν έχει τεράστιες ε, φιλοδοξίες για τους στόχους του 2020, αλλά η χρηματοδότηση αυτών των προγραμμάτων και των στρατηγικών αντιμετωπίζουν πάρα πολλές περικοπές. Άποψή μου είναι ότι υπάρχει ασυνέπεια. Πώς μπορείτε να αναγκάσετε την ε, Κομισιόν να αφιερώσει περισσότερα κονδύλια για το 2013 για το έτος Ιθαγένειας και για το ζήτημα του φίλου Αν δεν έχετε χρήμα δεν μπορείτε να πετύχετε φιλόδοξους στόχους. Και κάτι ακόμα ερωτώ. Εντάξει, θα σταματήσω εδώ. Πώς ε, μπορείτε να ζητήσετε περισσότερη χρηματοδότηση για τις πολιτικές ισότητας ε, και τα σχετικά προγράμματα και να αυξηθεί το ποσό από ένα εκατομμύριο στο ποσό που είχε δαπανηθεί στο παρελθόν, λαμβάνοντας υπόψη ότι θα έχουμε και εκλογές ευρωπαϊκές το 2014 και θέλουμε να εκλεγούν περισσότερες γυναίκες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κλάση. Ευχαριστώ πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ τη Δανική Προεδρία για την παρουσία της εδώ. Έχω στην Επιτροπή Περιβάλλοντος αυτές τις μέρες. Είδα Υπουργό της, ε, του Περιβάλλοντος, είδα Υπουργό Γεωργίας, είδα Υπουργό ε, Υγείας τώρα ε, και τον Υπουργό για θέματα γυναικών. Μεγάλη χαρά λοιπόν συναντώ τη Δανική Προεδρία και πιστεύω ότι μπορούμε πολύ από την Ευρώπη να διδαχθούμε από αυτά που γίνονται στο βορρά της Ευρώπης για να ισχύσουν σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πιστεύω θα είναι καλό παράδειγμα. Και πιστεύω ότι έτσι έχετε και την ευκαιρία να διαδώσετε αυτή την αντιμετώπιση σε ολόκληρη την Ευρώπη. για τις παρατηρήσεις ότι η Γερμανία τίνει μάλλον προς την εξοικονόμηση πόρων. Θα ήθελα να συμπληρώσω ότι και στον χώρο της, ε, τον κοινωνικό δεν μπορούμε να έχουμε ε, ως μόνη λύση την πολιτική της εξοικονόμησης πόρων γιατί αν θέλουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους πάνω απ' όλα θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να μπουν στον χώρο της εργασίας και ως εκ τούτου δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε την οικονομία από την κοινωνία, από τα κοινωνικά θέματα δηλαδή. Ε, αυτό πρέπει πάντα να αποτελεί μια γενική αρχή. Για την κυρία Φρέντριξεν, κυρία Υπουργέ, μιλήσατε για την Ευρωπαϊκή ημέρα για ισότιμη αμοιβή ότι θέλετε να ανακηρύξετε μια Ευρωπαϊκή ημέρα. Τι εννοείτε συγκεκριμένα και πώς μπορεί, εάν μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμμετάσχει και να συμπράξει αυτό. Εν γέννη, πιστεύω ότι η ισότητα μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο εάν συμμετάσχουν και οι άνδρες στην αγώνα αυτών. Ερωτώ λοιπόν τι έχετε υπόψη και οι δύο Υπουργοί. Στον κοινωνικό τομέα, στον επαγγελματικό χώρο, πώς μπορούν οι άντρες να συμπράξουν για το σκοπό της ισότητας και για την κυρία Φρέντριξεν πάλι σε αυτό που είπατε ότι η κρίση πρέπει να αντιμετωπιστεί σαν ευκαιρία και να την αξιοποιήσουμε. Ναι, αυτό νομίζω ισχύει για ολόκληρη την Ευρώπη. Και αν ε, θέλουμε να στρέψουμε το βλέμμα προς το μέλλον, πρέπει να διαπιστώσουμε ότι γυράσκει ο πληθυσμός μας, η κοινωνία μας. Στην ε, Γερμανία, παραδείγματι, έχουμε ήδη έλλειμμα σε νέους ε, που θα μπορούσαν να αναζητήσουν κατάρτιση δεν υπάρχουν αρκετοί νέοι δηλαδή που να πηγαίνουν σε εξειδίκευση, σε μαθήματα κατάρτιση, ενώ στην ε, Ισπανία Φερρυπίνη η κοινωνία είναι πολύ πιο νεαρή. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να πάψει η Γερμανία αυτό που κάνει, αλλά να αναπτύξει μια συνεργασία για ένα κοινό πρόγραμμα ε, εκπαίδευσης και επαγγελματική κατάρτισης που να επιτρέπει και στους νέους να αξιοποιούν τις δυνατότητες που υπάρχουν σε κάποια άλλη χώρα. Γιατί ο Ισπανός νέος να μην είναι σε θέση να πάει σε ένα άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να λάβει μια καλή εκπαίδευση κατάρτιση επαγγελματική που θα του είναι χρήσιμη ε, πιστεύω ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις εθνικές δομές και πολλά άλλα κοινωνική ε, συνεργασία σε κοινωνικά θέματα και να εξασφαλίσουμε χάρη στην εργασία αυτή μια Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ καλύτερα εξοπλισμένη για να αντιμετωπίσει μεγάλες προκλήσεις στο μέλλον. Και αυτό θα πρέπει να αφορά τόσο άνδρες όσο και γυναίκες. Πρέπει πάντοτε να θέτουμε το θέμα αυτό υπό την έννοια της ε, Συμμετοχή πεστρών γυναικών στον χώρο εργασία και τη μείωση τη ενέργεια. Ευχαριστώ πολύ. Actually, uh... Πρόεδρε, ευχαριστώ. Πρέπει να σημειώσω ότι ήδη γνώριζα την, ε, το πρόγραμμα της Δανικής Προεδρίας γιατί πριν από μερικές εβδομάδες συναντηθήκαμε στην Κοπενχάγη και ήδη πρέπει να πω ότι με εντυπωσιάσατε. το γεγονός ότι τέτοια χώρα έχει αναλάβει την ε, ηγεσία τώρα και την καθοδήγηση συζήτηση αποτελεί για μένα εγγύηση ότι θα προχωρήσουμε πολύ καλά και πολύ γρήγορα. Ε, κάτι το οποίο υπόθηκε όμως ιδιαίτερα και επαναλήφθηκε αρκετέ φορές, δεν ήθελα να υπογραμμίσω, το θέμα της άδειας μητρότητας. Το πρόβλημα που έχουμε τώρα είναι ότι έχουμε τη γρομοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του άμεσα εκλεγμένου θεσμικού όργανου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία παρακολύουν κάποια ε, μέλη του Συμβουλίου, κάποια μέλη του Συμβουλίου, δεν καν ολόκληρο το Συμβούλιο. Και γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να βάλουμε πάνω απ' όλα τη δημοκρατία, πάνω απ' όλα να βάλουμε στι σωστέ διαστάσει σωστές διαστάσεις όλη αυτή τη συζήτηση. Και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι οποιαδήποτε τέτοια θέματα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε με δημοκρατία και με δημοκρατική υπευθυνότητα. Νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρη υπουργό το θέμα αυτό. Βεβαίω θέλουμε τη διαδικασία της διαλλαγής αν το προτιμάτε ή κάποια άλλη τέτοια προσέγγιση. προς τις θέσεις του Συμβουλίου οι οποίες επιφυλάξει ενδεχομένω έχει, αλλά υπάρχουν κάποια βασικά ζητήματα. Διάρκεια μητρικής άδεια, πλήρης αποζημίωση και ευθύνη ή συνυπευθυνότητα του πατρός, δηλαδή συμμετοχή και του πατέρα στην, ε, σε ένα βαθμό κατά κάποιο τρόπο στην μετρική άδεια. Βέβαια ξέρω ότι, πολλά κρατημέ... ότι κάποια κρατημέλη έχουν πάρα πολύ σκληρή στάση στην υπόθεση αυτή. Ξέρω ότι η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου είναι επίσης πολύ σκληριστική στη θέση, αλλά νομίζω ότι πρέπει να συνεργαστούμε για να καταλήξουμε σε καλές θέσεις, θετικές θέσεις στο θέμα αυτό. Επίσης, άλλο ένα θέμα που θέλω να σας προτείνω, να σας υποβάλω. Υπάρχει μια νέα έκθεση που το κανονισμό για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εκεί βλέπω ένα σημείο. Διαδική προσέγγιση ε, κατά τρόπο προαιρετικό και όχι υποχρεωτικό. Αυτό νομίζω ότι αντιβαίνει στις βασικές αρχές και για την ισότητα των ανδρών και γυναικών και ε, σε άλλα θέματα, σε άλλες βασικές αρχές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω ποιε ε, είναι, Ποιε είναι οι απόψει στο θέμα αυτό εν τέλει. Κυρία Κυρνίλσεν το ανέφερε νωρίτερα. Η κρίση η διέξοδος από την κρίση κατά τρόπο οικονομικό αλλά και περιβαλλοντικό θα πρέπει να έχει μια προσέγγιση με βάση την ισότητα των φύλων. Δεν μπορούμε να ε, προφασιστούμε την κρίση για να αναβάλουμε την υλοποίηση των μέτρων ε, για ισότητα των ανδρών και γυναικών ε, που έχουμε ήδη αποφασίσει στο παρελθόν των αντίων, Πρέπει να τα υλοποιήσουμε και κατά πιο ουσιαστικό ακόμη τρόπο. Γιατί μέχρι στιγμή δεν είναι ουσιαστική και δεν είναι αποτελεσματική και ικανοποιητική η εφαρμογή του. Και νομίζω ότι η δική σα κυβέρνηση είναι η καταλληλότερη για να ηγηθεί αυτή τη προσπάθεια. Σα διαβεβαιώ από πλευρά των πρασίνων τη Ευρώπη ότι θα έχετε την υποστήριξή μα. Καλώς, ευχαριστώ πολύ. Κυρία Λούρινγκ έχει το λόγο. τελευταία Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη που έφτασα με καθυστέρηση. Ζητώ συγγνώμη και από τους εκπροσώπους της Δανεικής Προεδρίας. Βρισκόμουν σε μια άλλη συνεδρίαση. Μου είπαν όμως ότι συζητήθηκε το ζήτημα της οδηγίας σχετικά με την ε, αδιαμητρότητας ε, που έχει μπλοκαριστεί στο Συμβούλιο να πω στο Δανική Προεδρία ότι κατανοώ απόλυτα την θέση του Συμβουλίου διότι δυστυχώς ε, και προειδοποίησαμε εμείς στο παρελθόν περί αυτού παραφορτώσαμε τη βάρκα ιδιαίτερα εδώ στην Επιτροπή μας και δυστυχώς ε, παρά αυτό το υπέρβαρο πετύχαμε μια πλειοψηφία στο Νολομέλη διότι ουδής είχε το θάρρος να πει ανοιχτά ότι με μια παρόμοια έκθεση δεν έχουμε καμία δυνατότητα, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πετύχουμε τον στόχο της ε, άδειας μητρότητας που επιθυμούσαμε εάν δεν είχαμε παραφορτώσει το ε, σκάφος είμαι σίγουρη ότι η οδηγία σχετική με την προστασία της μητρότητας ε, θα είχε προοδεύσει, ίσως όχι σημαντικά, αλλά μια κάποια πρόοδος θα είχε επιτευχθεί κάτι που είναι σημαντικό για τα κράτη-μέλη που ακόμα βρίσκονται στο κατώτατο όριο της της οδηγίας. Δεν μπορούμε να τα αναμειγνύουμε όλα σε μια οδηγία Γι' αυτό και το Συμβούλιο δεν ξέρει τι να κάνει με την έκθεση αυτή. Γι' αυτό σας είπα ότι καταλαβαίνει το Συμβούλιο. Εμείς δεν είμαστε κατά βελτίωσης ε, των των επιπέδων προστασίας της μητρότητας, αλλά στην πολιτική πρέπει πάντα να γνωρίζουμε τι είναι εφικτό και τι όχι. Ε, η Ισπανική Προεδρία προετών μου είχε πει ότι αν υιοθετήσετε την έκθεση αυτή υπό την σημερινή μορφή να το ξεχάσετε. Δεν πρόκειται να προχωρήσει διότι ξεπερνάει τις κόκκινες γραμμές. Θέλουμε να βελτιώσουμε την προστασία της μητρότητας ή ε, άδεια πατρότητα είναι άλλο πράγμα, η άδεια άλλο. Αλλά εάν τα μπλέξουμε όλα μαζί, φίρδιν μίγδιν, καταλαβαίνετε ότι δεν θα οδηγηθούμε πουθενά. Ο Ταϊλεράνδος είναι αυτός που είπε ότι οτιδήποτε είναι υπερβολικό δεν έχει ουσία, δεν έχει έννοια, δεν έχει νόημα. Και εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο αυτό πράξαμε. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στους υπουργούς σου. και μετά θα κάνω κάποια τελικά σχόλια. Θα στεγώ κάποια συμπεράσματα. Ποιος θέλει να ξεκινήσει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για τα ευγενικά σας λόγια. Δεν έχω συνηθίσει σε τέτοιες αυρότητε. Σα ευχαριστώ πάντω για τη συζήτηση. Νομίζω ότι αυτό αποτελεί και την καλή προϋπόθεση για μια, συνεργασία, την για μια καλή συνεργασία. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούμε να προχωρήσουμε με βήμα αλλά <clears throat> ελπίζουμε ότι μια κάποια πρόοδος θα επιτευχθεί μήνα με το μήνα, χρόνο με το χρόνο. Ε, έγιναν ε, πολλά σχόλια σχετικά με την οδηγία περιμητρότητας και με ικανοποίηση έλαβα σήμερα μία επιστολή και μου άρεσαν τα σχόλια του κυρίου Ταραμπέλα για την ε, ανάγκη επίδειξης ε, ευελιξίας και πολλές φωνές ε, είπαν ότι επιθυμούν ένα πραγματικό διάλογο με το Συμβούλιο και επιθυμούν να αυτό που είπα και νωρίτερα. Δεν πρόκειται να εξυπηρετήσουμε κανενός ε, τα συμφέροντα εάν δεν προχωρήσουμε σε έναν διάλογο. Γι' αυτό λοιπόν θα φροντίσουμε αυτή η συνεργασία, αυτός ο διάλογος να λειτουργήσει ε, υπό δανεική Προεδρία και ενδεχόμενα να πετύχουμε κάποιο συμβιβασμό επί του περιεχομένου. Αλλά πρωτού φτάσουμε στο συμβιβασμό θα πρέπει να ξεκινήσουμε να... την συζήτηση, τη διαπραγμάτευση. Αυτό το οποίο επιθυμεί το Κοινοβούλιο, από ό,τι διακρίνω, είναι να βελτιωθούν ε, η κατάσταση σε θέματα ισότητας, ε, ισορροπίας ε, στο πλαίσιο της οδηγίας περιμητρότητας και όλα αυτά προς όφελος των κοινωνικών δικαιωμάτων. Το Συμβούλιο ε, θεωρώ ότι με ικανοποίηση θα καταγράψει μια τέτοια βούληση. Εσείς παράλληλα πρέπει να κατανοήσετε την πολιτική πραγματικότητα, ότι το Συμβούλιο θα πρέπει να πλοηγηθεί ανάμεσα σε αυτά τα 27 κράτη-μέλη και στις 27 θέσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις αμοιβές, ε, ξέρετε ότι αυτές ε, διαφέρουν από κράτος σε κράτος και σε ό,τι αφορά την ε, ρύθμισή τους. Υπάρχουν ουσιαστικέ πολιτικές διαφορές στο πλαίσιο του Συμβουλίου και επίσης σε ό,τι αφορά την ταχύτητα με την οποία μπορούμε να προοδεύσουμε. Αλλά πρέπει να κατανοήσουμε τι βρίσκεται πίσω από τις προθέσεις του Συμβουλίου, πίσω από τις προθέσεις του Κοινοβουλίου. Αυτά θα μας επιτρέψουν τουλάχιστον να ξεκινήσουμε να εργαζόμαστε προς την αυτή κατεύθυνση και ενδεχόμενα να καταλήξουν σε ένα συμβιβασμό. Κάτι που άκουσα με ικανοποίηση ότι και εσείς επιθυμείτε. Και γι' αυτό σας ευχαριστώ. Τώρα, για το active aging, για την ενεργό ηλικία, δηλαδή με τα, από ποια ηλικία οι γυναίκες μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται. Ε, στο, στην ε, συνάντηση της Κοπενχάγης ε, το συζητήσαμε το ζήτημα και το θέμα της ενεργού και επιθυμούμε οι άνθρωποι να δουλεύουν περισσότερο το ζήτημα είναι κατά πόσον μπορούν να δουλέψουν μετά από κάποια, εργασία, κάποια ηλικία Αυτό φυσικά θα εξαρτηθεί και από την αγορά εργασία ε, τώρα. Ε, ε εάν ε, δεν έχετε κάποια ειδίκευση, μετά από τα 65-70 είναι πολύ δύσκολο να παραμείνετε στην αγορά εργασία. Εκτό αν έχετε ε, κάποια πτυχία, κάποια διπλώματα που σας επιτρέπουν να εργαστείτε σε άλλες εργασίες, όχι σκληρές κλπ. Αλλά ε, αυτό που μας ενδιαφέρει και μας ε, ως ε, Δανική Προεδρία είναι να βελτιωθούν οι δεξιότητες και τα προσόντα των πολιτών. Το, το ζήτημα της ένδυας και το θέμα της δεξιοδότησης πρέπει λοιπόν να βελτιώσουμε την ε, κατάσταση των γυναικών στον χώρο της εργασίας, στην απασχόληση. Αυτό νομίζω ένας, είναι ένας στόχος στον οποίο όλοι, ε, στον οποίο όλοι ε, συμφωνούμε, αλλά πρέπει να εξετάσουμε πώς μπορούμε να το πετύχουμε. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το θέμα των ε, βρεφονιμπιακών σταθμών ε, είναι πολύ σημαντικό. Εάν ε, μπορούμε να έχουμε μια ημερήσια φροντίδα υψηλής ποιότητας, τότε οι γυναίκες δεν θα χρειαστεί να εγκαταλείψουν την αγορά εργασίας, διότι δεν θα χρειαστεί να ασχοληθούν αποκλειστικά με τα τέκνα τους. Και κάτι ακόμα. Χαίρομαι που ακούω αυτές τις υψηλές προσδοκίες που τρέφεται για την Ιδανική Προεδρία. Πάντως ε, σας υπόσχομαι ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Και βλέπω ότι η Προεδρία δεν είναι μόνη της. Αν μπορούμε να συνεχίσουμε λοιπόν αυτήν την συνεργασία μεταξύ ημών και ημών σίγουρα θα πετύχουμε πολλά, σε υπόψη και την περίοδο κρίση την οποία διανύουμε. Ευχαριστώ. Για είναι με σπισέτη σύστη Συμφωνώ απόλυτα με την ε, συνάδελφο. Ναι, αλλά να απαντήσω σε κάποια ερωτήματα κ. Μέου μίλησε για το κοινωνικό ταμείο και τις ε, διαπραγματεύσεις επί του νέου κανονισμού που αφορά το κοινωνικό ταμείο το 2013-2020. Δεν είμαι εγώ άμεσα αρμόδιος για το ζήτημα, αλλά στο Συμβούλιο επιθυμούν να πετύχουν μια κοινή θέση, κάτι που θα αποτελέσει ε, μια βάση για περαιτέρω συνεργασίες, ε, συζητήσεις με το Κοινοβούλιο. Τώρα σε ό,τι φορά τα ποσοστά, το Συμβούλιο συμφωνεί με την ε, ισότιμη συμμετοχή ανδρών και γυναικών σε όλα τα επίπεδα και χρειάζεται να είμαστε θέση να χρησιμοποιήσουμε και να υποφέρουμε από όλες τις δεξιότητες, όλες τις, όλα τα προσόντα που διαθέτει η Ευρώπη. Το Συμβούλιο υποστηρίζει την ίση συμμετοχή των γυναικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και πρόκειται να προτείνει μέτρα για να αυξήσει τον αριθμό των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια που θα συζητηθεί στο, υπό την ε, Δανική Προεδρία. Και ξέρουμε ότι θα γίνει μια συζήτηση στις 17 Φεβρουαρίου στο Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ για την υποεκπροσώπηση γυναικών σε διοικητικές θέσεις. και αυτά φυσικά θα ε, διαβαστούν στην ε, Κομισιόν. Τώρα, η ε, συνάδελφός μου είπε και αυτή ότι πρέπει να προχωρήσουμε, πρέπει να αναλάβουμε κάποια, να κάνουμε κάποια βήματα. Και τώρα, σε όλη φορά την κυρία να σας ευχαριστήσω για τα καλά σας λόγια, για την υποστήριξη και ευχαριστώ και τον κύριο Ταραμπέλα. Το mainstreaming είναι φυσικά απαραίτητο για την πρόθεση της ισότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε σχέση με τις κλιματικές αλλαγές και το ζήτημα των μεταφορών. Ε, όλες οι αρχές ε, θα πρέπει να λάβουν υπόψη το θέμα της ισότητας ε, των φύλων. Αυτό φυσικά απαιτεί να έχουμε και θέσεις οι οποίες θα στηρίζονται σε στατιστικές, σε στοιχεία, σε δεδομένα. Θέλουμε λοιπόν μια πολύ καλή βάση. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την ε, σημερινή συζήτηση. Αγαπητά μέλη του Κοινοβουλίου, αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ με... και είμαι βέβαιος ότι μιλώ και εξ ονόματος της συναδέλφου αποτέλεσε ιδιαίτερη χαρά που βρεθήκαμε σήμερα ανάμεσά μας σας διότι αυτό συμβαίνει άπαξ στον βίο μας σε 13 χρόνια θα ξανά έχει η Δανία την Προεδρία και δεν ξέρω αν σε 13 χρόνια αφενός ε, θα ζω και αφετέρου αν θα έχω ακόμα αυτό, κατέχω ακόμα αυτό το θόκο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Υπουργέ. Ε, παρακαλώ, καθίστε, μη μιλάτε. Θα ήθελα να κλείσω τη συζήτηση αυτή λέγοντας ότι εγώ δεν υπέβαλα ερωτήσεις προς τους υπουργούς επειδή είχαμε τόσο μακρύ κατάλογο μιλητών και ήθελα όλοι οι άλλοι να μπορούν να υποβάλουν τις δικές ερωτήσεις. Κυρίως όμως ε, θα ήθελα να πω ότι έχω ήδη συναντήσει δύο φορές και τους δύο υπουργούς και μπόρεσα να συζητήσω μαζί τους αυτά τόσο σημαντικά θέμα. Βασιζόμενος λοιπόν στην θέση της, ε, του Κοινοβουλίου υπέβαλα τις ερωτήσεις που ήταν για μας σημαντικές. Σας παρακαλώ λίγη ησυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, όταν συνάντησα τον Υπουργό κ. Σαρίνε, ένα από τα πιο σημαντικά θέματα που συζητήσαμε ήταν η στάση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη βία κατά των γυναικών και τη στρατηγική που θέλουμε να ακολουθήσουμε όταν συζητιώνται τα θέματα αυτά για να μην έχουμε κατακαιρματισμένη στάση. Και με την Υπουργό κ. Φρέντεντιξεν συζητήσαμε προφανώς για το θέμα της σημασίας της ε, Άδεια μητρότητα. και χάρηκα που η Υπουργό Φεντερικσέν θέλει να κάνει ό,τι μπορεί στο τομέα αυτό και ο Υπουργό Σαρίν ό,τι μπορεί στο δικό του τομέα. Και χαίρομαι που η ε, Δανική Προεδρία θεωρεί ότι και το θέμα του περιβάλλοντος και του κλίματος είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, γιατί ξέρετε ότι υπάρχουν και άλλα θέματα που συζητήσαμε που δεν είναι θέμα μόνο όντως άνδρων και γυναικών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμο για όλους που μπορούσαν να συζητήσουν τα θέματα αυτά τόσο επικοδομητικά. Η υπουργό ε, κυρία Φιντερίξεν είπε «Α, πολύ καιρό μας διαθέτεται, πολύ χρόνο μας διαθέτεται γι' αυτό». Και είπα «Ναι, αλλά η δική μας επιτροπή χαίρεται να υπάρχει συζήτηση και να ε, υποβάλει ερωτήσεις και να ακούει τις απαντήσεις. Καταλάβατε λοιπόν γιατί έγινε αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

with the committee meeting and Okay. Uh, uh, hello everybody. Ε, do so... Λοιπόν, σας παρακαλώ. Όποιος θέλει παρακαλώ να κουβεντιάσει. Ευχαρίστως να το κάνει απ' έξω από την αίθουσα, γιατί πρέπει να αρχίσουμε να ψηφίζουμε. Επαναλαμβάνω, ποιος θέλει να έχει συνομιλίε κατηδίαν, εκτός τη αίθουσα, παρακαλώ. Εμείς πρέπει να αρχίσουμε εδώ τώρα με την ψηφοφορία, τις ψηφοφορίες. Λοιπόν, περνάμε τώρα στο σημείο 13. και θα δώσω καταρχήν το λόγο στην κυρία Κένεν. Ευχαριστώ πάρα πολύ Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις πολιτικές ομάδες, ιδίως τους κοιόδες ηγητές που συνεργάστηκαν πάρα πολύ, επικοδηματικά και καλά μαζί μου. Και να σας ευχαριστήσω και για την υπομονή που δείξατε και τις ικανότητες να επιτευχθεί συμβιβασμό. Πριν από την ψηφοφορία θα ήθελα να επιστρέψω την προσοχή σας σε δύο σημεία. Καταρχήν, υπήρχαν ε, γλωσσικές δυσκολίες σε αυτό το κείμενο. Καμιά φορά να βρεθεί η σωστή διατύπωση για κάποιες από τις ε, τροπολογίες. για να μπορούν να είναι σύμφωνα με τις εκάστοτε εθνικές ε, εκλογικές νομοθεσίες. Σε ορισμένε χώρες υπάρχει δυνατότητα ποσοστώσεων, σε άλλες όχι. Λοιπόν, υπάρχουν αυτές οι συμβαστικές τροπολογίες, μπορείτε να τις διαβάσετε. Ό,τι επιτρέπουν τις πολιτικές ομάδες. Έχω τη συμφωνία των Δημοκρατών, Άλτε και Πρασίνων. και παρόλο που ήταν τις τελευταίες στιγμές πέτυχα να έχω στα χέρια μας τις επιλογές. Μετά στον ε, κατάλογο ψηφοφορίας μπροστά σας βλέπετε τις ε, προφορικές τροπολογίες που έχουν συμφωνηθεί. Δεν πρόκειται να τις διαβάσω όλες, θα τις βρείτε στο κείμενο. Και σας λέω, έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Σας ευχαριστώ όλους λοιπόν για άλλη μια φορά. και ελπίζω μετά την ψηφοφορία και τη συμφωνία θα μπορέσουμε να συζητήσουμε πώς θα προωθήσουμε το περιεχόμενο της έκθεσης. Με συγχωρείτε, τεχνικό θέμα. Δεν θέλω να ψηφίσω, αλλά έχει σπάσει η κάρτα μου. Μπορείτε να με μετρήσετε συμπληρωματικά. Ναι, δύο άτομα πρέπει να μετράμε. Έξτρα. Κοιτάξτε, εγώ την ξέχασα, δεν μου την έσπασα, την κάρτα μου. Α, ευτυχώς, ευτυχώς οι συνεργάτες μου είναι αποτελεσματικοί και μόλις μου έδωσαν την κάρτα που είχα ξεχάσει. Okay. Πολύ ωραία. Θα αρχίσουμε λοιπόν την ψηφοφορία. Συμβαστική τροπολογία 2. Ποιο είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Οι 35, 34, 33, 37 και 36 καταπίπτουν λοιπόν. Και περνάμε στην συμβασική τροπολογία 3. Ποιος είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Αν κρίνεται επίσης ξεκάθαρα. Οι 38 και 39 καταπίπτουν λοιπόν. Ψηφίζουμε την τροπολογία 40. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 41. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. κρίνεται. τροπολογία 4. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται ξεκάθαρα 48, 46, 43, 47, 45, 44, 42 και 49 καταπίπτουν λοιπόν και περνάμε στη συμβασική τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 56, 59, 58, 54, 55, 53, 50, 52, 57 και 51 κατά πίπτων. Και ψηφίζουμε την... Όχι την εξή, θα την ψηφίσουμε αργότερα. Συμβαστική 6. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Οι 61 και οι 72 καταπίπτουν λοιπόν. Και περνάμε στην τροπολογία 62. Υπέρ, κατά, αποχές. Για να το ελέγξουμε αυτό. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 62 άρχεται. Πέρας πληροφορίας. 13 συν 2, 15 υπέρ δηλαδή και 16 κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 63. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 65. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρι... συγγνώμη. Να ελέγξουμε, να ελέγξουμε, ευχαρίστω. 65, να ελέγξουμε την 65. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Το ΕΛΚ έχει μία ψήφα παραπάνω από ό,τι δικαιούται. Τώρα εντάξει. Πέρασε ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 16 προς 16. Τροπολογία 64. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 66. Με μια προφορική τροπολογία. Ψηφίζουμε και την προφορική τροπολογία. Ωραία, δεν είναι κανένας αντίθετος. Ψηφίζουμε λοιπόν. Είσαστε κατά τη προφορικής. Α, περνάμε λοιπόν στην, στην τροπολογία χωρίς αυτό. Ποιος είναι υπέρ. Στην επιτροπή μόνο ένας αρκεί. Λοιπόν, ψηφίζουμε την τροπολογία 66, αρχική. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Άποχες. Για να ελέγξουμε. Την αρχική τροπολογία 66. αρχή ψηφοφορία. Πέρας. Στο ΕΡΤ υπάρχουν ε, περισσότεροι ψηφίζοντες από ό,τι δικαιούνται. Με την κυρία Κράτσα δύο παραπάνω έχουμε. Τώρα εντάξει. Τώρα εντάξει. Τώρα είμαστε εντάξει. Λοιπόν, 16 προς 15 και μία εποχή Εγκρίνεται. Με μία ψήφο πλειοψηφία. Οι δύο που ψηφίζουν ε, με ανάθεση χειρός ε, ψηφίσαν υπέρ, γι' αυτό εγκρίνεται. Είναι 14 συν 2. Τροπολογία 67. Όχι, 69 υπέρ. Α, όχι, όχι, όχι, όχι. Ναι, ναι, πραγματικά έπρεπε να ψηφίσουμε 67. Ναι, ναι, ναι, ναι, σωστά. Και με μία προφορική τροπολογία είσαστε κατά. Ωραία. Λοιπόν, ψηφίζουμε την αρχική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ της 67, παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 69. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Άρα πρέπει να ψηφίσουμε τις 68. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 70 καταπίπτει. 71. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 72 έχει καταπέσει και το 76 το ίδιο 74 λοιπόν υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίθηκε νομίζω 73 έχει ήρθε η 75 καταπίπτει επίσης γιατί 74 είναι νεκρήθη συμβαστική τροπολογία 8 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται άρα οι τροπολογία 77, 78, 80 καταπίπτουν Συμβαστική 14 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Οι 82, 79, 80 και 81 καταπίπτουν λοιπόν. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Οι 84, 85 και 86, 87 και 83 καταπίπτουν. Τροπολογία 88. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ροδανέα καταπίπτει. Ενενήντα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. ένα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 92 έχει καταπέσει. 95 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 94 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 93 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Να ελέγξουμε την 93 παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Το ΕΛΚΑ έχει έναν περισσότερο από τους δικαιούται ψήφους. Απορρίπτεται. Τροπολογία 96. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Για να ελέγξουμε. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 96 παρακαλώ. Άρχισε ψηφοφορία. Okay. The vote is closed. Πέρασε. Εγκρίνεται ξεκάθαρα. 97 καταπίπτει. 98 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 99 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 100 έχει καταπέσει. 101 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 102 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Την 102 θέλετε να ελέγξουμε. Εντάξει. Να ελέγξουμε την 102 ηλεκτρονικά. Missing one. The vote is closed. It's rejected. Απορρίπτεται. Συμβαστική 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άρα 103 και οι 60 καταπίπτουν. Συμβαστική 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Οι 105 και 106 καταπίπτουν. 108, 107 και 104 καταπίπτουν. 109 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται να ελέγξουμε η 109 άρχιτη ψηφορία πέρασε. Απορρίπτεται. 113 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 112 απεσύρθη 111 λοιπόν 111 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. Να ελέγξουμε την 111. Άρχιτε ψηφοφορία. The vote is closed. Πέρας. Απορρίπτεται. Πρόβλημα. Το μηχανάκι δεν δουλεύει. Ψηφίζω όχι και βγαίνει αποχή. μόλις πάντησα όχι και ε, γράφεται ως αποχή. Έτσι με καταχωρεί. Λοιπόν, ε, τότε να μας δείχνετε με ένα της χειρός για να σας καταμετρήσουμε αν έχετε προβλήματα. Όχι, όχι. Το, το πράσινο δεν λειτουργεί, το κόκκινο δεν λειτουργεί. Δεν θα άλλαζε τίποτα για αυτή τη διαδικασία όμως, για αυτό το γύρο. Sorry, it's... Okay. Uh, we, we want to. Uh, those are in favor on one. Λοιπόν, 110 υπέρ. Κατά. Αποχές. Για να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για την 110. Πέρασε πληροφορίες. Ξεκάθαρα είναι κρίθη. Τροπολογία 114 καταπίπτει. Ψηφίζουμε τα 115 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 116 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 117 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 118 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 119 καταπίπτει 120 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρα 121, 122, 123 και η 131 καταπίπτουν. Περνάμε στην 126. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 125. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 127 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 124 έχει καταπέσει και 128 επίση. ψηφίζουμε λοιπόν το 130 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 129 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 131 έχει καταπέσει 132 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και μετά έχουμε στην τελευταία αυτή σκέψη μια προφορική προσθήκη Τη ΕΡΠΑ Πιετήκεν, της ηγήτριας. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 9. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 10. Υπέρ, κατά, απόχέ, εγκρίνεται. Τροπολογία 11. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 με μια προφορική τροπολογία. Τη δεχόσαστε? Όχι, δεν τη δεχόσαστε. Αρχική λοιπόν τροπολογία. 16. Έχει τροπολογία 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβέχει τροπολογία 1 Μήπω ε, δεν είδα καλά και είπα 11. 1 εννοούσα. Λοιπόν, τροπολογία 1. βασική τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Οι 19, 20 και 21 καταπίπτουν. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Οι 24 και 25 λοιπόν καταπίπτουν. Και περνάμε στην τροπολογία 26. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 28. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 27. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 29. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αυτό σημαίνει 31 και 32 καταπίπτουν. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. με αναφορά 7 με μια προφορική τροπολογία. Διαφωνεί κάποιος με την προφορική τροπολογία. Δεν εκπλήτωμε ότι διαφωνείτε. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σέβομαι το δικαίωμα να είναι κανένα αντίθετο με τι προφορικέ τροπολογίε αλλά αυτό δεν ε, προσθέτει κάποιο περιεχόμενο απλώς αναφέρεται στη σωστή μορφή της απόφασης ε, του Ηνωμένων Εθνών. Είναι τεχνικής μορφής δηλαδή αυτή η τροπολογία. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι πρόκειται για πολιτική δήλωση με το οποία είμαι Και έχω το δικαίωμα να το κάνω. Και θέλω να σας πω ότι στην Ολομέλεια υπέβαλα μια πολύ σημαντική ε, προφορική τροπολογία για τα δικαιώματα των κρατουμένων, στο οποίο ανετάχθη το ΕΛΚΑ. Πρόεδρος, όχι, όχι, έχει το δικαίωμα να είσαι αντίθετος. Δεν κατάλαβα τι συζητάμε αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται να συζητάμε. Α, έχει το δικαίωμα να απορρίψει μια προφορική τροπολογία. Αυτοί είναι οι κανόνες. Λοιπόν, προχωράμε στην τροπολογία 2. Κύριε Παπανόφ, με συγχωρείτε. Αν δεν το αλλάξουμε με προφορική τροπολογία, θα έχουμε ψηφίσει το λάθος ψήφισμα. Δηλαδή τι εικόνα θα παρουσιάσουμε προς τα έξω. Παραδέχομαι το δικαίωμα του συναδελφού, αλλά είναι τεχνικής μορφής αυτό, αυτή η τροπολογία. Πρόεδρος, κοιτάξτε. Εμείς τώρα δεν ε, μπορούμε να συζητήσουμε την διαδικασία. Όποιος θέλει αυτή η τροπολογία να περάσει θα πρέπει να την υποβάλει σαν τροπολογία στην Ολομέλεια. Δεν είναι τόσο τραγικό. Έτσι νομίζω. Λοιπόν, άλλο το διαδικαστικό και άλλο το πολιτικό. Το διαδικαστικό είναι σαφέ. Περνάμε τώρα στην οπλογία 2. Υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και στο σύνολο του ψηφίσματος η ηλεκτρονική ψηφοφορία η οποία άρχεται τώρα πέρασε ψηφοφορίας Προσθέτουμε τις δύο βέβαια. 26 προς 3 και 2 αποχές. Λοιπόν, εγκρίνεται η πρόταση. Συγχαρητήρια κύριε Πίτικεν. And now we're moving on to... Και τώρα περνάμε στο επόμενο σημείο. Απαλληλή 2010, Γενικό Προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυρία Ματέρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι συνεργάστηκαν για την κατάρτιση αυτών των δύο νομοδοτήσεων. Εύχομαι η Επιτροπή Προϋπολογισμών που συνεδρίασε σήμερα και θα συνεδριάσει και στο μέλλον να επικεντρωθεί στις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου αλλά και στα θέματα που αφορούν την Επιτροπή μας διότι στο παρελθόν δυστυχώς έγιναν πολλές περικοπές και αυτές οι περικοπές έπεσαν στο κεφάλι μας. Ελπίζω λοιπόν στο μέλλον να έχουμε έναν προϋπολογισμό πολύ πιο ισχυρό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορούμε λοιπόν να περάσουμε στην ψηφοφορία της πρότασης. Παράγραφος 2, τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται ξεκάθαρα. Στην παράγραφο 3 υπάρχει μια τεχνική διόρθωση, δεν θα την ψηφίσουμε. Τροπολογία 2 όμως. Ποιο είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά παρακαλώ. Για το σύνολο του ψηφίσματος. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. 25 προς 3. Εγκρίνεται λοιπόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ την εισηγήτρια. Και περνάμε στην δεύτερη έκθεση της κυρίας Ματέρα. Θα ξέρω να της ξαναδώσω το λόγο. Θέλετε το λόγο κυρία Ματέρα. Όχι. Εντάξει. Μπορούμε να περάσουμε εμείς την ψηφοφορία. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθη νομίζω, για να ελέγξουμε. Ε, έπρεπε να το πω εκ μιας αρχής βέβαια. Άρχιψη ψηφορία για την τροπολογία υπεριθμών 1. Πέρας. Ναι, ναι, είναι κρίθη πράγματι. Τροπολογία 2. Υπέρ. Α, όχι, έχει καταπέσει, συγγνώμη. Ναι, ναι, έχετε δίκιο. Τροπολογία 3. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. Να ελέγξουμε, ευχαρίστω. Στην τροπολογία παρελθόν 3. Πέρας. Ενεκρίθη. Τροπολογία 4 για 4. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία για το κείμενο. Άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ευχαριστώ κυρία Ματέρα για μια φορά. We now moving on and uh, if you please could. Uh, Ας προχωρήσουμε τώρα παρακαλώ. και αν θέλετε να αποχωρήσετε παρακαλώ ησύχως για να συνεχίσουμε τη συνεδρίαση. Και μια και τέλειωσε η ψηφοφορία, ξαναρχίζω με τα σουηδικά μου. Συνεχίζω λοιπόν και γυρνάμε στα Σουηδικά παρακαλώ. Κυρίε και κύριοι, ναι και τέλειωσαν οι ψηφοφορίε. Περνάμε στο σημείο 14. Εξυγχρονισμό των συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και δίνω το λόγο αμέσως στην κυρία Τσέσκοβα, εισηγήτρια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον εισηγητή ε, επί της ουσίας από την Επιτροπή Πολιτισμού και Εκπαίδευσης που ετοίμασε την έκθεση αυτή να κάνω την παρουσίασή μου. Θα ήθελα να στήσω συγγνώμη από τους σκιώδεις συγγητές Γιατί ε, μου ανακοινώθηκε ότι θα πρέπει να αναλάβω τη γνωμοδότηση αυτή πολύ πρόσφατα, την προηγούμενη εβδομάδα, στο Στρασβούργο. Και χρειάστηκε να εργαστώ πολύ βιαστικά. Δεν ε, μπόρεσε λοιπόν να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής μας μέχρι και σήμερα ακόμη η μεταφρασμένη έκδοση της γνωμοδότης αυτής. Αλλά η πίεση χρόνου οφείλεται στο γεγονός ότι πρέπει ή θέλει η Επιτροπή Πολιτισμού και ε, Εκπαίδευση να, ε, και Παιδείας να ψηφίσει το ταχύτερο δυνατό την κύρια έκθεση. Ελπίζω λοιπόν ότι θα έχουμε την ευκαιρία αργότερα να συστήσουμε διεξοδικά τα θέματα με τους κοιόδης οδησηγητές. Κάποιες γενικές παρατηρήσεις λοιπόν για την ε, γνωμοδότηση. για να σα εξηγήσω τι ήταν, ποιοι ήταν οι λόγοι τους, οι οποίοι με υποχρέωσαν να συμπεριλάβω τις παρατηρήσεις μου στην, ε, στο κείμενο. Φυσικά και η εκπαίδευση έχει πολύ μεγάλη σημασία για την ανάπτυξη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια έχουν ακόμη τεράστιο δυναμικό το οποίο δεν αξιοποιείται επαρκώς στο πρόγραμμα 2.14.2020 ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα συζητήσουμε μάλιστα σήμερα ακόμη προτείνεται ε, ο προπολογισμό για τι επενδύσει στην ε, εκπαίδευση, την έρευνα να αυξηθεί και γι' αυτό πρέπει να συζητήσουμε τα θέματα αυτά. Είναι πολύ κοντά βέβαια σε θέματα μιας έκθεση που συζητήσαμε πρόσφατα για, τις, ε, για την παρουσία των γυναικών στην έρευνα και την επιστήμη. Ίσως λοιπόν να ε, δούμε κάποιες επαναλήψεις πράγματα που έχουμε ήδη συζητήσει σχετικά με την έρευνα και την επιστήμη. Για να επανέλθω στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, προτείνεται ο εξυγχρονισμός των ευρωπαϊκών συστημάτων, ε, των πανεπιστημιακών συστημάτων της εκπαίδευσης. Θα ήθελα να υπογραμμίσω τα συστήματα, το πρόγραμμα Εράσμου, το οποίο έχει διευκολύνει ιδιαίτερο τις ανταλλαγές φοιτητών, και που θεωρώ ότι αποτελεί μια πολύ καλή πρόταση και προϋπόθεση για επιτυχία στην αγορά εργασίας των νέων αυτή η δυνατότητα ανταλλαγών. Πρέπει λοιπόν να τίνουμε προς, μια, προς ένα υψηλότερο επίπεδο ανώτατης εκπαίδευσης και να αξιοποιούμε όσο δυνατόν περισσότερο το δυναμικό που υπάρχει. Στην ομοδότησή μου επικεντρώνομαι σε θέματα που θεωρώ σημαντικά. Η παρουσία των γυναικών σε πανεπιστημιακούς κύκλους αυξάνεται, ναι, αλλά δεν είναι επαρκής ε, η εκπροσώπηση των γυναικών ε, σε, σε συγκεκριμένου τομεί ε, και αυτό νομίζω οφείλεται και σε ιστορικούς λόγους και παραδοσιακές πεπιθήσεις περί ε, διάκρισης ε, μεταξύ των φύλων, περί παραδοσιακών ρόλων των φύλων. Αυτό ε, αντικατοπτρίζεται και στα, στο πανεπιστημιακό χώρο και στην επιλογή του πεδίου μάθησης των φύλων. Φαίνεται ότι στις θετικές επιστήμες δεν εκδηλώνουν ενδιαφέρον συχνά οι γυναίκες, οι νεαρές γυναίκες. Και ίσως αυτή η προσέγγιση σε μεγάλο βαθμό να οφείλεται σε παραδοσιακά, παραδοσιακές νομοτροπίες. Έτσι λοιπόν είναι πολύ πιο δύσκολο ε, οι γυναίκες να βρεθούν σε ισότιμη ανταγωνιστική βάση με τους άντρες για την αγορά εργασίας. Το έχει να κάνει και με τη συμμετοχή στην έρευνα και την επιστήμη. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι θα πρέπει να είναι περισσότερη η εκπροσώπηση των γυναικών στην, ε, στα ε, σώματα, στα κέντρα λήψης αποφάσεων και για τα πανεπιστήμια. Πολλές φορές όταν ε, λαμβάνεται μια απόφαση για την ανάθεση ενός ε, μιας υψηλής βαθμίδας ε, εκπαιδευτικής σε άντρα ή γυναίκα, η απόφαση αυτή δεν είναι ουδέτερη και μερόληπτη. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσία των γυναικών. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα βέβαια που αντιμετωπίζουν στον δρόμο τους οι γυναίκες. Πολλές φορές για λόγους των οικογενειακών τους υποχρεώσεων διακόπτουν τη σταδιοδρομία τους η γυναίκα. Αυτό βέβαια επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο εάν και οι δύο ε, σύντροφοι και οι δύο σύζυγοι ε, προέρχονται από τον χώρο των πανεπιστημίων, οι καθηγητές. Πρέπει να βρεθούν λύσεις, να δοθούν λύσεις οι οποίες θα ε, εξασφαλίζουν ισότιμη στήριξη του επαγγελματικού επιστημονικού βίου και του οικογενειακού και έτσι πιστεύω μπορούμε να έχουμε ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και υποψηφίους ύψης του επίπεδου, εάν καταφέρουμε να τα συγκεράσουμε αυτά. Παραλαμβάνω ε, κλείνοντα ότι είχα πολύ λίγο χρόνο για να προετοιμάσω τη γνωμοδότησή μου και πραγματικά περιμένω με αδημονία τις προτάσεις ε, υποδείξεις των συναδέλφων για να τις συμπεριλάβω στο κείμενο. Ευχαριστώ πολύ. Eh, Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Κυρία Παλιαδέλη. Το μικρόφωνο σας είναι κλειστό. Well, uh, I read it with interest. Μελέτησα με ενδιαφέρον την ε, γνωμοδότηση και ευχαριστώ την συγκεκριά, τη συντάκτρια για την δουλειά που έκανε σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Θα ήθελα να σημειώσω δύο παρατηρήσεις για το σημείο Β. B. Εκεί που αναφέρεται ότι αναφέρονται οι χώρες στις οποίες είναι περιορισμένος ο αριθμός των γυναικών που συμμετέχουν σε κέντρα λήψη αποφάσεων. Δεν θα ήθελα ρητή αναφορά. Θα ήθελα να διαγραφούν δηλαδή τα ονόματα των κρατών. να υποστηρίξουμε βέβαια την ιδέα, αλλά να τροποποιηθεί η διατύπωση. Και αυτό είναι μόνο μία πρόταση βέβαια, εσείς θα το κρίνετε. Θα σας καταθέσω μια τροπολογία και κρίνετε εσείς. Συμφωνώ πλήρως με τα περισσότερα επόμενα, με τα άρθρα. Στο σημείο 3 έχω κάποιες επιφυλάξεις. Αντιλαμβάνομαι ποια είναι η προσέγγιση σας, αλλά η πρόταση να αναθεωρηθούν τα κριτήρια για προαγωγή σε ανώτερες ερευνητικές θέσεις. Δεν νομίζω ότι αρμόζει σε γυναίκες που έχουν αγωνιστεί ε, σε ισότιμη βάση και έχουν καταφέρει να γίνουν καθηγητές. Τις υποδομές τα κατηγορούσα εγώ περισσότερο. Τις υποδομές που δεν μας επιτρέπουν να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, να διεκδικήσουμε ισότιμα κριτήρια, δηλαδή αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια. Θα έλεγα λοιπόν ότι πρέπει το σημείο αυτό να επαναδιατυπωθεί τελείω. Γιατί δεν την ότι από ίκτο προσφέρουμε κάποια ευνοϊκή μεταχείριση στις γυναίκες. ή ζητάμε από τους άντρε να δείξουν κατανόηση γιατί οι γυναίκε έχουν και άλλες υποχρεώσεις. Κριτήρια ισότιμα λοιπόν. Αλλά να υποστηρίξουμε με άλλο τρόπο την ε, αναρρίξη των γυναικών στην ιεραρχική ε, πυραμίδα, στα πανεπιστήμια, όχι γιατί είναι γυναίκες, αλλά γιατί ε, έχουν τα, την επάρκεια την επιστημονική που απαιτεί ο κάθε κλάδος. Κατά τα άλλα συμφωνώ, αλλά θα ήθελα να συμπεριλάβω μια αναφορά στη δυνατότητα για ε, ομάδες, μάλλον ε, εκπροσώπους μειονοτήτων όπως Φερρυπίν ε, και πρόσφυγες ε, να ε, εντάσσονται σε προγράμματα γλώσσας, κατάρτισης κτλ. Δηλαδή και προγράμματα ε, διαβίου μάθησης εν γέννη. Επίσης θα με ενδιαφέρει να συμπεριληφθεί μια αναφορά σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο να, ενταχθεί στα προγράμματα σπουδών των πανεπιστημίων ειδικό μάθημα για την ισότητα των φίλων. Σε αυτά όλα συμφωνώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλει κάποιος άλλος να λάβει το λόγο παρακαλώ. Αν όχι... Ας απαντήσει η κυρία Τσέσκοβα αν θέλει. Ναι, με συγχωρείτε ένα λεπτό. Η Επιτροπή βεβαίως. Σέντεν. Η μία από τις δύο θέλει να λάβει το λόγο. Έχουμε κάποιον εκπρόσωπο από την Επιτροπή να λάβει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί πολύ σημαντική τη διάσταση της, ε, του φύλου, της ότιμης του φύλου, όπως άλλωστε καταγράφεται και στην ανακοίνωση Σεπτεμβρίου και ιδιαίτερα όσον αφορά τις ευκαιρίες για μια γυναίκα να προχωρήσει, να αναρριχηθεί σε υψηλότερα κλιμάκια της ε, ιεραρχικής ε, πυραμίδας στα πανεπιστήμια, στον χώρο τη της Ευχαριστώ πολύ. Καλώς, λέει ο πρόεδρος. Τώρα η συγκήτρια. Και πάλι. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο και βέβαια ευχαριστώ και για τα σχόλια. Ασφαλώς θα φροντίσω να συμπεριληφθούν στις τροπολογίες, ε, με τις τροπολογίες, σα μάλλον στο κείμενο και με τον τρόπο αυτό να βελτιώσω όσο μπορώ το κείμενο. Για το τελευταίο σχόλιο της Επιτροπής, θα ήθελα να σημειώσω απλώς ότι μου φαίνεται πολύ σαφές, πολύ σαφής η τοποθέτηση της Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ. Eh, λοιπόν, τότε σημειώνουμε το χρονοδιάγραμμα. Παρακαλώ για την πρόταση κατάθεση τροπολογιών μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου. ψηφοφορία στην Επιτροπή 27-28, Επιτροπή Πολιτισμού 29 Φεβρουαρίου, Ολομέλεια τον Απρίλιο. Ωραία, έτσι έκλεισε και αυτό το θέμα και πάμε στο υπαριθμό 15. ετήσια έκθεση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα να τον κόσμο κατά το 2009 και την πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση επί του θέματο συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων για τη στρατηγική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέτρο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Well, this is a ε, opinion of the... Πρόκειται για ένα σχέδιο γνωμοδότηση και νομίζω πως ε, Αρχικά η έκθεση ήταν για το 2010, αλλά άλλαξε η ημερομηνία και έτσι μπορούμε να λάβουμε υπόψη ε, κάποια γεγονότα του 2009. αλλά και το 2011, διότι η ημερομηνία τελικά είναι το 2012. Θα σας ε, πω τι ακριβώς ε, πιστεύω. Τώρα στη γενική προσέγγιση μιλάω για διακρίσεις κατά γυναικών. Αναφέρω ότι ε, αυτό δεν μπορεί να δικαιολογηθεί για κανέναν πολιτιστικό, πολιτισμικό ή θρησκευτικό λόγο. Η βία κατά των ε, γυναικών θεωρώ ότι είναι κάτι το είδε χθες όπως επίσης και η κακοποίηση παιδιών, γυναικών που εξακολουθεί να ασκείται, να ασκείται ως, ε, με τρόπο μάλλον απαράδεκτο. Οι γυναίκες διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην ε, μεταπολιματική προσπάθεια για οικοδόμηση της ειρήνης, ε, επίλυση συγκρούσεων, συμφιλίωση και αποκατάσταση. Πρέπει να αναγνωρίσουμε λοιπόν αυτόν τον ρόλο στις γυναίκες. Ειδικά θα ήθελα να υπογραμμίσω την ασφάλεια των παιδιών, ειδικά των γυναικών στον τρίτο κόσμο. Διότι συχνά πέφτουν θύματα κακοποίησης και βιασμών. Εν, τώρα. Επίσης, να αναφερθώ στο ρόλο των Ηνωμένων Εθνών ε, στην υποστασία των ε, δικαιωμάτων της γυναίκας και καλούμε την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τοποθετήσει το ζήτημα δικαιωμάτων γυναικών στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων με υποψήφιε προ ένταξη χώρε. Επίση, αναφέρομαι για τι επαναστάσει στην Αίγυπτο, τη Λιβύη, την Τινησία, την λεγόμενη Αραβική Άνοιξη διότι οι γυναίκες διαδραμάτισαν πολύ σημαντικό ρόλο για την ελευθερία και για τα δικαιώματα των ε, κοριζιών και των ε, γυναικών. Η έκθεση ε, είπα ότι αφορά στο 2011, αλλά θα μπορέσουμε συνάμα να συμπεριλάβουμε και γεγονότα του 2011 όπως τα επανάσταση στις αραβικές χώρες. Επίσης με ανησυχεί το ζήτημα ε, των γάμων που γίνονται σε πολύ μικρές ηλικίε. Είναι, έχουμε οικογένειες οι οποίες ε, στέλνουν τα κορίτσια τους ε, στην Ευρώπη, μόλις ότι έχουν μεγαλώσει σε χώρες όπως η Ισία, η Ινδία κλπ. για να παντρευτούν μεγαλύτερους. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε κάτι για να αποφύγουμε αυτούς τους καταναγκαστικούς γάμους ε, και τη σεξουαλική βία και την σωματεμπορία. Έχουμε το ευρωπαϊκό, έχουμε τη σύμβαση για την εξάλληψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γενικών, αλλά έχουμε και το ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, αναφέρουμε επίσης στα δικαιώματα των γυναικών στην Τουρκία. Ε, το, μας απασχολεί ιδιαίτερα και ζητάμε από την Κομισιόν να ε, ζητήσει από την Τουρκία να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της και απαιτείται να επιδείξει εμφανή και από τα αποτελέσματα σε την εφαρμογή της αρχής ισότητας. Επίσης ε, ζητάω να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τα βραβεία Ζαχάροφ και ιδιαίτερα αυτά που έχουν ε, απονεμηθεί στις ε, γυναίκες. Αναφέρομαι επίσης στην επιλεκτική άμβλωση. Ε, κάποιες χώρες όπως η Κίνα και άλλες που εφαρμόζουν την επιλεκτική άμβλωση όταν η γυναίκα περιμένει κορίτσι τότε επιλέγει να προχωρήσει σε άμβλωση. Συζήτησα προχθές με τους κοιόδης ηγητές, μου είπαν ότι έχουν κάποιες ιδέες σχετικά με υποβολή τροπολογιών. Θα δω τι θα μπορέσω να κάνω προκειμένου να βελτιώσω περαιτέρω την γνωμοδότηση αυτή. Αν επιθυμείτε μπορώ να σας δώσω το λόγο. Κύριε Παπαδοπούλου, έχει το λόγο. Να κάνω μια σύντομη παρέμβαση δήλωσε. Είμαι σιώδης εισηγήτρια των σοσιαλιστών. Νομίζω ότι αυτή η γνωμοδότηση καλύπτει όλες τις ανάγκες των γυναικών σε αφορά τα δικαιώματά του στον τρίτο κόσμο, καλύπτει θέματα σώματα εμπορία, σεξουαλική κατοποίηση και άλλε μορφέ διακρίσεων. Έχει μεγάλη σημασία η Ευρωπαϊκή Ένωση και η στρατηγική τη ανθρώπινα δικαιώματα να αντανακλάται στην νομοθεσία τρίτων χωρών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να δραματίσει σημαντικό ρόλο για την συμπερίληψη πολιτικών που αφορούν στην ισότητα των φύλων και να ξεπεραστούν τα εμπόδια και φραγμοί που υπάρχουν σε διάφορους τομείς της, υγεία, της ε, ζωής. Εγώ προσωπικά προτίθεμαι να καταθέσω τροπολογίες. Η μία θα αφορά το γεγονό ότι στην Τουρκία παρά το, τις, ε, τις πολλές αλλαγές που έχουν γίνει ε, οι διακρίσεις κατά των γυναικών συνεχίζουν να υφίστανται παραβιάζονται τα, τα δικαιώματα των γυναικών και όταν ε, μεταβαίνουμε στην Τουρκία συζητάμε με μη κυβερνικές οργανώσεις και οργανώσεις γυναικείες που παραπονιόνται. Θα θέλαμε λοιπόν να συμπεριληφθεί αυτό στην παράφο 5. Σε ό,τι αφορά τους στόχους της χιλιετίας θα θέλαμε να ε, αναφερθούμε στην εφαρμογή αυτών των στόχων διότι η πρόοδος είναι πολύ αργή ειδικά σε ζητήματα που αφορούν την ε, ε, αναπαραγωγική υγεία. Ε, αυτές είναι οι πιο σημαντικές τροπολογίες, αυτά είναι οι πιο σημαντικά ζητήματα που, στα οποία θα εστιάσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μέντες, ε, θέλετε να λάβετε το λόγο πάλι να απαντήσετε. Ξέχασα να σα πω ότι η καταληκτική προθεσμία είναι η Δευτέρα Φεβρουαρίου για την υποβολή τροπολογιών και θα εξεταστεί ε, στις 27 και στις 28 Φεβρουαρίου η έκθεση ομού με τις τροπολογίες. Επειδή και εγώ είμαι σκιώδης και είχαμε χθες την συνάντηση των σκιωδών, και φυσικά ένα μεγάλο κομμάτι υποστηρίζει την γνωμοδότηση και η αναπαραγωγική υγεία και για των μητέρων είναι σημαντική. Να πω ότι η γνωμοδότησή σας είναι εξαιρετική. Το λόγο έχει η κυρία Uh, Ο κύριος, συγγνώμη. Ονομάζομαι Σπον και είμαι από την Υπηρεσία Δράσης. Ένα σύντομο σχόλιο ε, σχετικά με την γνωμοδότηση που βρίσκεται οποίο μας. Καλύπτει μια σειρά σημαντικών ζητημάτων. Είναι ένα πεδίο όπου συνεχώς λαμβάνουμε καλές ειδήσει. Ε, είπατε πρόσωπος ε, φρόντισε να προωθήσει τα δικαιώματα των γυναικών και να καταστήσει προτεραιότητα. Υπάρχει και ένα κείμενο το οποίο τώρα βρίσκεται στα σκαριά. Τώρα για το κείμενο που έχουμε αναχείρασα ασχολείται με την ετήσια έκθεση του 2010. Αλλά η γνωμοδότηση ούτε στα εκτιμώνες ούτε στις πολλέ παραγράφου σου κάνει αναφορά στην ετήσια έκθεση και Διαρωτώ με πώς βλέπει τη σχέση μεταξύ αυτής της ε, νομοδότησης και την εργασία του κ. Χάβορντ. Να δώσω τώρα το λόγο στην εισηγήτρια κυρία Χιμένες. Ε, ε, Μου ενημέρωσαν πως η έκθεση έφτασε με καθυστερημένα και είχαμε συμφωνήσει ότι δεν θα λάβουμε αναφορά στο 2010 Γι' αυτό το λόγο λοιπόν θέσαμε και το θέμα της Αραβικής Άνοιξης διότι είχαμε πει ότι δεν θα γίνει χρονική αναφορά στο 2010 επειδή έφτασε με καθυστέρηση η έκθεση αυτή. Και μια που πρόκειται να υποβληθεί η γνωμοδοσία του 2012, προτιμήσαμε να καλύψουμε και ένα κομμάτι του 2011 αν και δεν θα ήταν σωστό να μιλήσουμε για μέχρι και το 2010, γι' αυτό προτιμήσαμε να μην βάλουμε την ημερομηνία του 2010, διότι προχωρήσαμε στο 2011 εμείς. Λοιπόν, όπως είπε η κυρία Χιμένες, η καταληκτική ημερομηνία κατά της τροπολογιών είναι η Δευτέρα Φεβρουαρίου και θα ψηφίσουμε στις 27 και 28. Η ΑΦΕΤ θα ψηφίσει τον Μάρτιο και στην Ολομέλεια θα πάμε τον Μάιο. Απρίλιο, συγγνώμη. Επόμενη συγγήτρια δεν βρίσκεται μεταξύ μας προς το παρόν καθοδόν είναι. Περιμένουμε λοιπόν λίγα λεπτά. Λυπούμε, αλλά περιμένουμε λίγο, γιατί είναι καθοδόν η συγχύτρια. Θα έρθει πολύ σύντομα στην αίθουσα. Okay, we continue and I... Λέω να συνεχίσουμε. Προλάβατε να πάρετε μια ανάσα. Ζητώ συγγνώμη, συγγνώμη που σας ε, πιέζω. Κύριε Ζούμπερ, να λάβετε λόγο λοιπόν. Καταρχήν, ζητώ συγγνώμη. Ε, ότι το σε μια άλλη επιτροπή όπου έκανα ε, την παρουσίαση μιας έκθεσης. Θα αναφερθώ στο κείμενο εργασίας, στο το οποίο έχει καταρτήσει η κυρία Φιγκερέιδο σε ό,τι αφορά το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020. Λοιπόν, στις προτάσεις, στο έγγραφο αυτό θεωρούμε ότι η άποψη της Κομισιόν σε ό,τι αφορά το φύλλο δίνει μεγαλύτερη ευελιξία σε ό,τι αφορά τις μελλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες. Τώρα, στο έγγραφο εργασίας, κατά την άποψή μας, της Κομισιόν, απουσιάζει μια δημοσιονομική πρικοδότηση θα έλεγα που θα αφορά τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων. Ναι, εντάξει, προβλέπονται κάποια κονδύλια για τους οριζόντιους στόχους, αλλά χρειάζεται να υπάρχουν και συγκεκριμένοι πόροι για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων. Υπάρχουν λοιπόν δύο επίπεδα, ένα εξειδικευμένο και ένα οριζόντιο, τα οποία θα πρέπει να είναι συμπληρωματικά μεταξύ τους. Και με πολλή ανησυχία παρατηρούμε ότι το αριθμό των εξοικειμένων μέσων όπως το πρόγραμμα Δάφνη περιορίζεται, μειώνεται. Το πρόγραμμα για την αντιμετώπιση των, της βίας από τις γυναίκες αλλά και σε ό,τι αφορά την ισότητα των, φίλων στο πλαίσιο του προγράμματος του Progress. Όταν ε, λοιπόν διαγράφονται κάποια συγκεκριμένα κονδύλια, αυτά δυστυχώς δεν αναπληρούνται από άλλα. Σε ό,τι αφορά τώρα την πρόταση αναφορικά με το πολιετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 δεν αντανακλά την ε, υποχρέωση ε, συμπερίληψης κάποιων προγραμμάτων που αφορούν θέσπιση ειδικού προγράμματο, ορισμού ισότητα των φύλων, ειδική δέσμευση χρηματοδότηση κλπ. χρειάζεται να υπάρξει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για τα ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών στο πλαίσιο της ιστορικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έπειτα στους ε, επιμέρους κανονισμούς θα πρέπει να αναφέρεται η ισότητα των φύλων ως συγκεκριμένος στόχος τόσο σε ό,τι φορά τους κανονισμούς των ταμείων αλλά και των προγραμμάτων. Επίσης ε, θα πρέπει να υπάρχει ειδική χρηματοδότηση στο πλαίσιο προγραμμάτων χρηματοδότησης και για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την ισότητα των φύλων. Λοιπόν, συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι η απόφαση του Συμβουλίου για το πολιετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένε ενδείξεις ε, και υποδείξεις προς την Κομισιόν με την συμπερίληψη των δικαιωμάτων γυναικών και της όρας των φίλων σε κάθε ένα από τα προγράμματα. Ένα από βασικούς δείκτες ε, σε ό,τι αφορά την τρόπο υλοποίησης ε, της χρηματοδότησης, όλα αυτά θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και την ε, επόμενη πενταετία Θεωρούμε λοιπόν πως χρειάζεται να καταρτιστεί ένα εξειδικημένο πρόγραμμα που θα αφορά αποκλειστικά τα... την ισότητα των φύλων που να έχει επίσης και μεγαλύτερη πορατότητα, μεγαλύτερη προβολή. Τώρα, σε ό,τι αφορά την χρηματοδότηση για τα ε, μη κυβερνητικές οργανώσεις και τα διάφορα έργα, τα διάφορα σχέδια. Ε, υπάρχουν ε, διάφορες ε, αλλαγές ε, που γίνονται και πολλά προγράμματα προωθούνται από τις μη κυβερνικέ οργανώσεις αλλά και από συνδικαλιστικές οργανώσεις προκειμένου οι μη κυβερνικές οργανώσεις να την χάνουν χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση οι επιδοτήσεις ίσονο σημασία θα πρέπει να συνεχίσουν να υπάρχουν παράλληλα με αυτές που αφορούν μεγαλύτερα ποσά. Επίσης, η χρηματοδότηση των μη κυβερνικών οργανισμών και της κοινωνίας των πολιτών θα πρέπει να είναι διαθέσιμα όχι μόνο για τα έργα, αλλά και να υποστηρίζουν την ανάγκη χρηματοδότησης της λειτουργίας και όχι μόνο χρηματοδότησης έργων. Τώρα, αναφορικά με το ζήτημα της ε, ηθαγένειας ε, θα πρέπει να συμπεριλάβουμε τον ε, στόχο και εδώ της ισότητας των φύλων. Θα πρέπει να προβλεφθεί και μια ελάχιστη χρηματοδότηση. Να, θα πρέπει να ενισχύσουμε περαιτέρω τις προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως το πρόγραμμα Δάφνη για να σταματήσει η βία κατά των γυναικών το ζήτημα του φύλου θα πρέπει να συμπεριληφθεί και στον Ευρωπαϊκό ε, για το Κοινωνικό Ταμείο και για την περιφερειακή ανάπτυξη που και οι θα πρέπει να συμπεριλάβουν τους στόχους της ισότητας των φύλων. Αυτά θα πρέπει να προκύψουν και από τα ειδικά ταμεία τα οποία αφορούν συγκεκριμένα προγράμματα όπως τα ευρωπαϊκά προγράμματα για την ισότητα, τη μετανάστευση, προγράμματα υγεία, ανάπτυξη, ορισμό 2020, ταμείο για το άσυλο κλπ. Πρόεδρο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει κανεί το λόγο. Κύριε Τσέσκου. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι συγκράτηση ηγέτρια και γι' αυτό έχω κάποια σχόλια να κάνω. Θα καταρχήν να ευχαριστήσω την συγκέντρια ε, μέσω ναι, ημών για αυτό που έκανα, για το έργο της. Ε, τα σχόλια μου αφορούν αυτά που είπατε. Γιατί πρόκειται για ιδέες που κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ κοντά είμαι με τις ΔΕ, από, όπως κρατώ την μου με μη κυβερνήσεις οργανώσεις. Παραδείγματος χάρη τα προγράμματα που υπήρχαν, Δάφνη, Progress, έχουν μειωθεί. Η σημασία του Δάφνη είναι διασυνδίτητη και η δική μας πολιτική ομάδα υποστήριζε αυτό το τομέα. Επίσης ε, θέλαμε να υπάρχει αύξηση του προπολογισμού του συγκεκριμένου ε, προγράμματος. γενικά νομίζω ότι θα πρέπει να υποστηρίζουμε τα προγράμματα τα οποία έχουν αποδειχθεί επιτυχή. Και ενδεχομένω να δούμε και περισσότερους πόρους. Αλλιώ, δεν πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στη σημερινή οικονομική κατάσταση θα πρέπει να κάνει κάτι διαφορετικό από την αύξηση των πόρων για την ισότητα των ε, φύλων, αλλά αυτό όμως εξοικονομώντα ε, πόρου από κάπου αλλού. Ας πούμε από προγράμματα που δεν ήταν επιτυχή. Στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού ξέρουν πολλού τέτοιου τομείς όπου τα προγράμματα δεν είναι επιτυχή. Οι πόροι που δίνονται στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Οργανισμό Ισότητα των Φύλων θα πρέπει να είναι επαρκή. Και εδώ αναφέρομαι στην πρόσληψη προσωπικού κάτι που θα ήθελα να τονίσω εκεί που λέγεται η χρηματοδότηση σχεδίων για τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις ε, υπήρχε μέλη για τις μικρές ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις οι οποίες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε μικρές ε, ποσότητες, σε μικρά ποσά χρηματικά στην μελλοντική χρηματοδοτική περίοδο θα πρέπει να μπορούμε να τους δώσουμε ακόμα μικρότερα ποσά για να μπορέσουμε να χρηματοδοτούμε πολύ περισσότερες από αυτές τις μικρές ε, μη κυβερνικές οργανώσεις γιατί πιστεύω ότι αυτές ακριβώς είναι εκείνες που είναι ο ακρογωνίος λίθος της ε, μάχης για την επίτευξη των στόχων μας. Τελευταίο σχόλιο η ισότητα των φυλών βασίζεται οπωσδήποτε στην οικογένεια, στα παιδιά αν θέλετε. Και γι' αυτό η παιδική στεθμή είναι κάτι που θα πρέπει να μας απασχολήσει. Ίσως να θέλουμε να το συμπεριλάβουμε στο έγγραφό μας. γιατί έτσι θα μπορέσουμε να υποστηρίξουμε αυτή την ιδέα ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ της εργασίας και της ε, ζωής ε, εκτός εργασίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει πρόεδρος. Θέλει κανένας άλλος να σχολιάσει. Υπάρχει κάποιος από την Κομισιόν εδώ που θέλει κάτι να πει επί του θέματος. Παρακαλώ. Πρόεδρε, θα κάνω ορισμένα γενικά σχόλια και μετά η Στάνφος μπορεί να προσθέσει ειδικά σχόλια για το πρόγραμμα που έχουμε μπροστά μας. Δεν να υπενθυμίσω ότι για την προετοιμασία των νέων ομοθετικών προτάσεων της Κομισιόν τα διάφορα αυτά προγράμματα είναι αντικείμενο μιας ε, ανάλυσης επιπτώσεων. Υπάρχουν κάποιες κατευθυντήριες γραμμέ. Ε, όσον αφορά τις επιπτώσεις στην, οικογένεια, στην κοινωνία και συγκεκριμένα στην ισορροπία ανδρών και γυναικών. Θέλω να σας πω ότι τα πιο σημαντικά προγράμματα και ενισότητα των φύλων είναι παραδείγματος οι πόροι που προβλέπονται στην πολιτική συνοχή. Οι νομοθετικές προτάσεις εδώ προβλέπουν ενδυνάμωση της λήψης υπόψη της ε, πολιτικής ισότητας. Παράδειγμα, η ισότητα ανδρών και γυναικών είναι μία τις οριζόντιες προϋποθέσεις για όλες τις προτάσεις μας στα πλαίσια του Δαμείου Συνοχής. Μια άλλη ενδιαφέρουσα πτυχή είναι ότι οι κοινέ διατάξεις ε, προβλέπουν τη λήψη υπόψη της ισότητας στην προετοιμασία και την εφαρμογή των προγραμμάτων. Αυτό είναι κάτι που ξεπερνάει αυτά που είχαν προβλεφθεί στην περασμένη ε, νομοθεσία. Και κάτι επίσης ότι το Οργανισμός για το Κοινωνικό Ταμείο προβλέπει όχι μόνο προγραμματισμό της λήψης υπόψη της ισότητας σε όλες τις παρεμβάσεις του, αλλά προβλέπει επίσης να συνοδεύει αυτό το gender mainstreaming με συγκεκριμένες δράσεις για να αυξήσει παραδείγματος χάρη την συμμετοχή των γυναικών στην πρόοδο, στην αγορά εργασία και στην απασχόληση. Και θα ήθελα να πω, για να τονίσω κάποια στιγμή τη έκθεση, ότι η ισότητα ανδρών και γυναικών λαμβάνεται υπόψη επίση και σε άλλα προγράμματα, παραδείγματο χάνει για τι κοινωνικέ αλληλεγγύε και την καινοτομία και στα προγράμματα τη έρευνα με τον Ρίζο 2020, καθώ επίση και στα προβλήματα για την υγεία. Αν μου επιτρέπετε, θα δώσω την συνάδελφο το λόγο για να συμπληρώσει τι πληροφορίε αυτέ. Ωραία. Πρόεδρε, όσον αφορά τα άλλα θέματα που θίγει η έκθεση. Καταρχήν, η έλλειψη συγκεκριμένων προγραμμάτων θα συνεχίσει στα αγγλικά μάλλον, όχι στα γαλλικά. Ο στόχος της Κομισιόν ήταν να μειωθεί ο αριθμός των προγραμμάτων, γιατί ακριβώς ο μεγάλος αριθμός προγραμμάτων το μία πηγή με παρκούς ε, διαχείρισης των ε, προγραμμάτων και επίσης προβλημάτων για τους δικαιούχους. Η Εγγύη Διεύθυνση για τη Δικαιοσύνη υπέβαλε επίσης ε, μια πρόταση για τα δικαιώματα των πολιτών όπου συμπεριλάβαμε το τέος πρόγραμμα Δάφνη και τις πτυχές ισότητας του προγράμματος Progress Δηλαδή το Δάφνη και το Progress δεν εξαφανίστηκαν, έχουν σωματωθεί σε ένα πιο ευρύ πρόγραμμα που συγκεντρώνει μια σειρά στόχων με στόχο να απλουστεύσει μεν, αλλά να μεγιστοποιήσει δε τις επιπτώσεις ε, της χρηματοδότησης. Στις προτάσεις αυτές ε, δεν προβλέψαμε προκαθορισμό χρηματοδότησης για συγκεκριμένους στόχους, όχι επειδή θέλουμε να εγκαταλείψουμε τη χρηματοδότηση θεμάτων δικαιωμάτων των γυναικών και ισότητας, αλλά για να έχουμε περισσότερη ευελιξία και να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα που υπάρχουν μακροπρόθεσμα, δηλαδή 2014-2020. Τέλος όσον αφορά τη χρηματοδότηση των μη κυβερνητικών οργανώσεων και των ε, προγραμμάτων τους. Το πρόγραμμα Δικαιώματα για τους πολίτες επιτρέπει την χορήγηση χρηματοδότησης σε μη κυβερνητικέ οργανώσεις στον τομέα της ισότητας των φύλων. Το μόνο πρόβλημα που έχουμε είναι ότι βρισκόμαστε εν μέσω οικονομικής κρίσης Και ο στόχος της Κομισιόν είναι να δώσει τα χρήματα εκεί που θα έχουν την μεγαλύτερη, το μεγαλύτερο αντίκτυπο. Και αναρωτιόμαστε πώς θα μπορούμε ιδανικά να πετύχουμε τους στόχους μας γενικά και τους στόχους της ισότητας των ε, φύλων. Κατά πόσο αυτό με το να χρηματοδοτούμε μικρές μη κυβερνικέ οργανώσεις ή αν αφήσουμε το θέμα αυτό στις εθνικές εξωτερικούς προπολογισμού, αυτό θα πρέπει να δούμε. Θα το εξετάσουμε μέσα στα πλαίσια του ετησίου προγράμματο ε, Πώ θα εφαρμοστεί δηλαδή. Και αυτό θα συζητηθεί με τα κράτη-μέλη και με το Κοινοβούλιο φυσικά. Αυτά σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και για να κλείσουμε η κυρία Ζούπερ. Πολύ γρήγορα. Θα ήθελα απλώ να σημειώσω ότι, να, να πω ότι σημειώνω Τι ερωτήσει που τέθησαν, σημειώνω τις παρατηρήσεις της κυρίας Τσέσκοβα και συνεχίζουμε τη δουλειά αυτή, λαμβανωμένων υπόψη των προτάσεων και παρατηρήσεων. Καλώς λέει ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ θερμά. Και έτσι κλείνουμε το σημείο 16, δηλαδή το τελευταίο σημείο της μέσης διάταξης, πάμε στο 17 στα διάφορα που δεν έχουμε τίποτα και στο 18 πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι αύριο έχουμε ένα σεμινάριο ή workshop για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα ξεκινήσουμε το πρωί στις 9 και ελπίζω ότι θα είστε όλοι και όλες παρόντες. Πρόκειται για την ε, προοπτική της όταση των φύλων στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Με μια κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής των, των Δημοσίων Ελευθεριών και της ε, Επιτροπής των Γυναικών που προβλέπεται για την επόμενη εβδομάδα για να συζητήσουμε την έκθεση για, ανθρώπινα, για τα δικαιώματα των γυναικών και η προσεχή συνεδρίαση εδώ προβλέπεται για τις 27 και 28 Φεβρουαρίου. Υπενθυμίζω ότι θα βρεθούμε αμέσως με τη λήξη συνεδρίασης ε, εδώ έξω στο διάδρομο για να πιούμε ένα ποτηράκι από χαιρετιστήριο καθώς η Σαμπίνε αποχωρεί, μας εγκαταλείπει. Θα της ευχηθούμε καλή τύχη και ευτυχία. Αυτό λοιπόν, αυτή η μικρή δεξίωση προς τη Μέντη Σαμπίνε θα λάβει χώρα εδώ ακριβώς έξω από την αίθουσα τώρα. Χαίρετε και ευχαριστώ